Καλησπέρα σας, καθίστε παρακαλώ. Καλημέρα ή καλησπέρα σε όλους σας. Είναι η πρώτη μας συνεδρίαση του 2014 και επ' ευκαιρία θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά. Κάπως καθυστερημένα, αλλά καλό αργά παρά ποτέ. Καλή χρονιά και πολύ καλή δουλειά. Ξεκινούμε με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Μήπως υπάρχουν αντιρρήσει για την ημερήσια διάταξη. Όχι. Δεν έχουμε λάβει καμία πρόταση για αλλαγή της ε, ημερήσιας διάταξης, οπότε θεωρείται ως συγκεκριμένη. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της 4ης και 5ης Νοεμβρίου και Δευτέρας Δεκεμβρίου 2013. Ε, τα πρακτικά αυτά σας έχουν μοιραστεί και αν έχετε σχόλια ως προς τα πρακτικά σας θέλω παρακαλώ να τα κοινοποιήσετε στη γραμματεία πριν το τέλος της απογευματινής μας συνεδρίασης. Αν δεν υποβληθούν ε, τροπολογίες ε, οι αντιρρήσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ε, τα πρακτικά θα θεωρηθούν ως εγκεκριμένα. Εντάξει. Έχουμε ανακοινώσει από την Επιτροπή. Ο λόγος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το κύριο Μακουάιτερ. Ελπίζω να προφέρω σωστά το όνομά σας. Ευχαριστώ. Δεν το προφέρατε και τέλεια, αλλά κατά προσέγγιση. Τρεις πρωτοβουλίες έχουμε για φέτος. Μία ανακοίνωση για την ενίσχυση του ρόλου του ιδιωτικού τομέα, για να έχουμε αηφόρο ανάπτυξη που θα περιλαμβάνει όλους και δεν θα αποκλείει κανέναν και θα δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις του ιδιωτικού τομέα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Θα έχουμε τη στρατηγική για την υλοποίηση του στόχου για το, το για την αλλαγή για ανάπτυξη χωρίς αποκλείς με ενεργό ανάμειξη του ιδιωτικού τομέα. Δεύτερον, έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών για την εφαρμογή των δεσμεύσεων που έχουμε αναλάβει σε θέματα επισητιστικής ασφάλειας η έκθεση αυτή θα θεθεί τον Ιούνιο και θα σας ενημερώσει για τις πολιτικές μας σε θέματα επιστημική ασφάλειας και ασφάλειας της διατροφής, καθώς και για τη γεωργία. Και θα έχουμε και την ετήσια έκθεσή μας, ως ήθιστε, για την ανάπτυξη των εξωτερικών μας πολιτικών και την εφαρμογή του για το 2013. Πέρυσι ολοκληρώθηκε το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα δούμε, θα κάνουμε ένα απολογισμό κατά το πέρας αυτού του δημοσιονομικού πλαισίου και θα αντλήσουμε κάποια συμπεράσματα από την εμπειρία μας. Αυτές είναι οι τρεις πρωτοβουλίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πρώτο εξάμεινο του 2014. Σας ευχαριστώ. Πολύ καλά. Περνάμε στην ώρα των ερωτήσεων. Έχουμε λάβει δύο ερωτήσεις για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρώτη είναι από τον κύριο Γκέρνς και έχει θέμα τον αντίκτυπο της διάσκεψης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου που έγινε στο Μπαλί και την αντίκτυπο στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η δεύτερη ερώτηση είναι της κυρίας Αργεντίνη και αφορά τις ποσοστώσεις για τη ζάχαρη. Σας έχουμε μοιράσει τις ερωτήσεις και θα ήθελα να παρακαλέσω τώρα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει πρώτα στην ερώτηση της κυρίας Αργεντίνη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα απαντήσουμε λοιπόν με την ευκαιρία αυτή στην ερώτηση. Είμαι διευθυντή ε, τη βιώσιμη ανάπτυξη στην σχετική, σχετική Γενική Διεύθυνση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζει την ερώτηση τη κυρία Σαρτζεντίνη η οποία μπορεί να επικεντρωθεί σε τέσσερι ε, άξονες. Η κατάσταση στο ότι αφορά την αγορά τη ζάχαρης μετά την μεταρρύθμιση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, ο αντίκτυπος ε, των μέτρων σε ό,τι αφορά τι στόχους της μεταρρύθμισης, οι προοπτικές ό,τι αφορά την εφαρμογή του MSP για να επιτρέψει την καλύτερη κατανομή των πόρων και επιπλέον χρηματοδότηση για την ε, διαφοροποίηση την οικονομική, μεταξύ άλλων και στρατηγικές για την διαφοροποίηση του κλάδου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υπενθυμίσει τα βήματα που οδήγησαν στην ε, κατάργηση των ποσοστώσεων στην ευρωπαϊκή αγορά ζάχαρης και την βοήθεια που έχει ήδη δοθεί στις χώρες ΑΚΕ για να ταπεξέλθουν στο νέο εμπορικό περιβάλλον. Το τέλος της παραγωγής ε, με ποσοστώσεις στον τομέα της ζάχαρης ήταν η τελική φάση που αποφασίστηκε το 2006, μια διαδικασία που αποφασίστηκε το 2006 και η αναθεώρηση του 2006, η μεταρρύθμιση, ε, περιλάμβανε ένα πακέτο 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ προς το AMSSP για να βοηθήσει τους σχετικούς παραγωγούς να ελαφρύνουν τον αντίκτυπο του 36% σε ό,τι αφορά τις ε, τιμές της ζάχαρης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αυξήσουν την αγωνιστικότητα και να βοηθήσουν τους άλλους παραγωγούς να διαφοροποιήσουν την παραγωγή τους. Και κάθε χώρα που επλήχθη ε, κατέστρωσε μια ξεχωριστή στρατηγική βάσει και των ξεχωριστών αναγκών της. Αυτό το γνωρίζω γιατί ήμουν επικεφαλής ε, της αντιπροσωπείας στα Φίτζη, στον Ειρηνικό, και το 2006 τα νησιά Φίτζη ανέπτυξαν μια ευρεία στρατηγική προς το σκοπό αυτό. Εξ αρχής λοιπόν ήταν σαφές ότι αυτή η αρρωγή θα ήταν προσωρινής φύσης και δεν θα έπρεπε να περιμένουν άλλη χρηματοδότηση πέρα από το 2013. Η εφαρμογή του μέσου θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις ξεχωριστές οικονομικές συμφωνίες και βάσει των αποφάσεων που περιλαμβάνονται στα μέσα αυτά πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ και 500 εκατομμύρια πρέπει ακόμα να καταβληθούν. Έχουμε λοιπόν ένα σχέδιο που μας βοηθά να καταλάβουμε την κατάσταση γιατί υπάρχει μια διαφορά μεταξύ της ανάθεσης και της καταβολής του ποσού. Και άρα δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί η διαδικασία σήμερα, θα συνεχίσει τα επόμενα χρόνια. Αυτή η εφαρμογή λοιπόν γίνεται με μία σειρά δράσεων. Και σκοπός είναι να υπάρχει ο μέγιστος δυνατός αντίκτυπος του μέσου. Αυτές οι δράσεις εξετάζονται τακτικά όπως προβλέπεται και στον κανονισμό. Και τα επιτεύγματα μεταξύ άλλων που έχουν ήδη επιτευχθεί είναι τα εξής. Σήμερα μπορούμε να αναφέρουμε ότι έχουμε ήδη σημειώσει κάποια επιτεύγματα προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση του 2006. Καταρχάς, οι εγκαταστάσεις έρευνας και οι σχετικές υπηρεσίες καταδεικνύουν ότι η προσαρμογή και τα σχετικά μέτρα για την προσαρμογή είχαν σημαντικό αντίκτυπο και στην ποιότητα αλλά και στην ποσότητα. Η Κένια, η Τανζανία, η Εκτή του και άλλες χώρες αποτελούν με ένα καλό παράδειγμα για αυτά. Κατά δεύτερον, οι μηχανισμοί για το δίκαιο εμπόριο έχουν συμβάλει στην βελτίωση του εργατικού, των εργατικών όρων. Σε κάποιες χώρες το βλέπουμε αυτό, όπως τα Φίτζη για παράδειγμα και στον Μπελιζέ. Και επεκτείνεται αυτά τα μέτρα και οι μηχανισμοί και στη Ζάμπια και στο Μαλάουι. Κατά τρίτον, η παραγωγή ζάχαρης και η μεταποίηση ζάχαρης ε, με πιο φιλικό προς, τον το περιβάλλον τρόπον ε, προωθούνται στην Τζαμέικα, στο Μαυρίκιο και το καθεξής. Επίσης, κάποιες χώρες μας απασχολούσαν ιδιαίτερως που αντιμετωπίζουν προβλήματα Τανζανία, Μαλάουι, ακτή του Ελεφαντοστού. Εκεί έχει βελτιωθεί η ο όγκος της ε, γεωργικής παραγωγής και προωθείται και ο διάλογος με άλλους συμπλεκόμενους φορείς όπως για παράδειγμα ο ίδιος ο κλάδος αλλά και οι σχετικές κυβερνήσεις στην Τζαμάικα και στην Κέινα. Κένια. Επίσης, ε, επέκταση των ε, υπηρεσιών που παρέχονται για να βελτιωθεί και η διαφάνεια μεταξύ άλλων. Τέλος, επενδύσεις σε συστήματα άρδρευσης. Αυτά προσέλκυσαν νέους ε, αγρότες στην αγορά αυτή και ενίσχυσαν και το κοινωνικό κεφάλαιο των παράγωγων, όπως για παράδειγμα στη Βοζαμβίκη και στη Σουαζιλάνδη. Αυτά λοιπόν είναι μεταξύ άλλων κάποια από τα παραδείγματα του αντικτύπου και συνεχίζουμε σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις ύψους 300 εκατομμυρίων και τα 500 εκατομμυρίων που πρέπει ακόμα να καταβληθούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρία Πρόεδρε, όπως και δεσμεύτηκε το 2013 για την τελευταία εκχώρηση τέτοιων πόρων, 100% των πόρων που είχε εκχωρήσει η χρηματοδοτική αρχή έχουν δεσμευτεί με ευέλικτο τρόπο εντός των ορίων που τίθενται από την νομική βάση. Για παράδειγμα, 60 εκατομμύρια πρόγραμμα για τα νησιά Φίτζη έχουν μεταφερθεί όμως σε άλλους δικαιούχους μετά από τα γνωστά επεισόδια και το πραξικόπημα το 2006 στα Φίτζι, καθώς ε, Υπάρχεται ακόμα στο άρθρο 96 η κυβέρνηση του Φίτζη σύμφωνα με την συμφωνία του Κοτονού και υπόκειται σε άμεση αρρωγή. Και έτσι λοιπόν αυτές οι δραστηριότητες παραγωγής της ζάχαρης ε, δεν εξαιρούνται από τα προγράμματα αυτά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο στη συμφωνία της, του Κοτονού αφιερώνουμε πάρα πολύ μεγάλο τμήμα στην ε, εταιρική σχέση, στην ιδιοκτησία. Άρα, αν η χώρα ζητήσει στα πλαίσια του προγραμματό να δράσει και να δραστηριοποιηθεί στον τομέα της ζάχαρης, είμαστε πολύ πρόθυμοι, όπως και σε άλλους τομείς της γεωργικής παραγωγής. Να πω ότι 49 χώρες, 49 χώρες έχουν ζητήσει την βοήθειά μας σε ό,τι αφορά τα προγράμματα ε, ασφάλειας τροφίμων, επιστικής ασφάλειας, γεωργικής παραγωγής και το καθεξής. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σε σχέση και με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο που μας είχε πιάσει κάπως απροετοίμαστος όταν σημειώθηκε η κρίση των τιμών των τροφίμων το 2008 και θυμάστε τότε τη διευκόλυνση για τα τρόφιμα που είχαμε διαπραγματευτεί από κοινού. Επιπλέον, η προσαρμογή της ε, ε, παραγωγής ζάχαρης ε, στις χώρες ΑΚΕ ήταν πιο ομαλή από ό,τι περιμέναμε. Και υπήρξε και σχετική έλλειψη στην ευρωπαϊκή αγορά. Οι ευρωπαϊκές τιμές λοιπόν δεν έπεσαν 36% όπως προβλεπόταν. Και έτσι η βάση της ε, συμφωνίας και της μεταρρύθμισης ε, είχε πάρει στο δεδομένο ότι θα έπεφτε η τιμή η παγκόσμια 36%. Δεν έγινε όμως αυτό. Σα το συγγνώμη κύριε Ριντόλφη. Ε, μπορείτε να, κατα... να ολοκληρώσετε γιατί έχουμε και άλλα θέματα και, άλλες... και άλλη ερώτηση. Και έτσι κατά συνέπεια λοιπόν, επειδή δεν έπεσε τόσο η τιμή, εμείς και η παραγωγή από τις χώρες ΑΚΕ καταφέραμε να προωθήσουμε τη ζάχαρη σε κερδοφόρες τιμές, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και αλλού. Και να πω ότι τέλος ότι ε, και ο ΣΑ και η ΦΑΟ προέβλεψαν ότι οι τιμέ της Ζάχαρη θα παραμείνουν υψηλέ στο μέλλον, πάνω από το μέσο όρο. Αλλά όταν έπεσαν ε, οι παγκόσμιες τιμές, η προνομιακή πρόσβαση στις χώρες Καριφόρμου θα ε, εγγυηθεί ένα πλεονέκτημα συγκριτικό και ανταγωνιστικό σε αυτές τις χώρες που θα διασφαλίσει ε, την οικονομική ευημερία στις χώρες αυτές, στις χώρες ΑΚΕ και στην Καραϊβική. Ευχαριστώ, λέει, κυρία Σαρχαντίνη, και ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πολύ εμπεριστατωμένη και εξονυχιστική απάντηση. Ελπίζω, αν την έχετε και γραπτός, να μας τη μοιράσετε. Υπάρχει εδώ μια διαφορετική αξιολόγηση, γιατί γνωρίζω ότι δεν είναι αναπάντεχο το τέλος του καθεστώτος της ζάχαρης, όλοι το περιμέναμε και μάλιστα μερικές χώρες, ε, η Νότια Αφρική, περιμένουν απεγνωσμένα αυτή την αλλαγή, γιατί δεν ανήκει στο καθεστώς ζάχαρη, Περιμένει πω και πώ το 2017 για να μπορέσει να διοχετεύσει το ζαχαροκάλαμό τη ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει όμως διαφορετική ερμηνεία μεταξύ ε, των χωρών ΑΚΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τι έχει γίνει και το πόσο έτοιμη είναι η, η κατάσταση. Πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε επανάληψη της περίπτωσης μπανάνας. Βέβαια, μπορεί να μας πει ο ΠΟΕ ότι δεν μπορεί να έχετε καλύτερη πρόσβαση στις μπανάνες των χωρών και σχέση με τις μπανάνες των χωρών της Λατινικής Αμερικής. Μήπως έχουμε κάτι αντίστοιχο. Και οι χώρες ΑΚΕ δεν ήταν ακόμη έτοιμες για κάτι τέτοιο. Τι κάναμε για να επιλύσουμε το πρόβλημα, περισσότερη ενίσχυση. Ε, είχαμε εμπορικές σχέσεις, αλλά χρειάστηκε να ενισχύσουμε την ε, συνδρομή προς τις χώρες ΑΚΕ. Ευχαριστώ για την εξήγηση αλλά δεν νομίζω ότι αρκεί αυτό για τις χώρες ΑΚΕ. Παρόλο που είναι αναμενόμενη η κατάσταση πέρυσι, οι χώρες ΑΚΕ, ή μάλλον 2012, είχαν πει οι χώρες ΑΚΕ σε μια διακήρυξή τους ότι δεν είναι ακόμη έτοιμες και φοβούνται την καταστροφή. Και μάλιστα ε, το αρμόδιο τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου πέρυσι τον Οκτώβριο δημοσίευσε μια έκθεση που έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για τις πιθανές δυσκολίες μιας τέτοιας ε, μετάβασης. Δεν νομίζω ότι λαμβάνεται υπόψη ο αντίκτυπος της ε, χώρας ΑΚΕ. Και παρά τις όλες προσπάθειες που μας εξεγγείλετε και που έχετε κάνει, πιστεύετε πραγματικά ότι οι χώρες ΑΚΕ είναι έτοιμες να δεχτούν την αλλαγή του καθεστώτος ή μήπως μπορούμε να κάνουμε και κάτι ακόμη. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ. Θα ξαναδώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσει στην ερώτηση του κυρίου Γκέρνς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είχα στείλει ένα ερώτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με τις τελευταίες διαπραγματεύσεις των ΠΟΕ στο Μπαλί και τον αντίκτυπο που είχαν στις ε, αναπτυσσόμενες χώρες. Θα θυμάστε ότι σε αυτό τον γύρο διαπραγματεύσεων, το βασικό θέμα ήταν και η ανάπτυξη μεταξύ άλλων. Κατά κύριο λόγο ήταν ένα γύρο διαπραγματεύσεων για την ανάπτυξη. Ποια είναι η αξιολόγηση λοιπόν τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ποιον αντίκτυπο είχαν οι διαπραγματεύσει αυτέ ή θα έχουν στι αναπτυσσόμενε χώρε, τι θα αλλάξει σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. Γνωρίζουμε ότι υπήρχε διαφορά απόψεων σημαντική με την Ινδία, άλλωστε και ο τύπο ασχολήθηκε με αυτό. Μπορείτε παρακαλώ να το σχολιάσετε πιο συγκεκριμένα. Και συν τη άλλη, αυτό που θα ήθελα να ξέρω τελικά είναι ποιος θα είναι ο αντίκτυπος ε, στον κλάδο της γεωργίας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Καλώς, θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στον κύριο Ζανσέλ Βανέκχοτ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον κύριο Γκέρενς για το ερώτημα αυτό. Είμαι επικεφαλής στις μονάδες για τις ε, διαθεσμικές σχέσεις, ε, διοργανικές σχέσεις στη Γενική Διεύθυνση για το Εμπόριο. Υπ' αυτή την έννοια ήμουν παρόν στο Παλί. Είχαμε σημαντική αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αποτέλεσε μέρος της επίσημης αντιπροσωπείας μας υπό τη διεύθυνση του καθηγητή κυρίου Μορέιρα διάσκεψη στο Παλί ήταν επιτυχημένη. Ήταν μια μέτρια επιτυχία, εάν δούμε το πόσο φιλόδοξη ήταν η στόχοι, πόσο μεγάλες οι φιλοδοξίες που είχαν τεθεί σε αυτό τον γύρο διαπραγματεύσεων το 2001. Ωστόσο παραμένει η επιτυχία. Γιατί, γιατί πρώτη φορά εδώ και πάρα πολλά χρόνια μια υπουργική διάσκεψη σε επίπεδο ΠΟΕ κατάφερε να καταλήξει εκεί που είχε σχεδιάσει, δηλαδή μια συμφωνία για τη διευκόλυνση του εμπορίου, αυτό είναι για πρώτη φορά από τη δημιουργία της σύσταση του ΠΟΕ. Για πρώτη φορά δηλαδή προστίθεται νέα συμφωνία στο υφιστάμενο σώμα συμφωνιών του ΠΟΕ και είχαμε και επιμέρους συμφωνίες για ε, πιο ίσονο σημασία ζητήματα, κυρίως ε, όσον αφορά στη γεωργία αλλά και στην ανάπτυξη. Να πω λοιπόν δύο λόγια για αυτά τα δύο καταρχάς. Ως προς τη γεωργία λοιπόν το βασικό ζήτημα το οποίο συζητήθηκε και επιλύθηκε στον Παλί είχε να κάνει με την επισητιστική ασφάλεια. Είχε τεθεί επιτάπητος από την Ινδία. Ειδικό πρόγραμμα, ούτως ώστε να υπάρχουν αποθέματα για να αντιμετωπιστούν καταστάσεις ξηρασίας ή λοιμού. Περιπτώσεις κατά τις οποίες η σοδιά δεν θα έφτανε για να θρέψει τον πληθυσμό. Αυτό το σύστημα λοιπόν ε, αντιβαίνει στους κανόνες του ΠΟΕ για τις εγχώριες επιδοτήσεις και ενισχύσει. Άρα ε, συμφωνήσαμε στον Παλί ότι προς το παρόν η Ινδία μπορεί να συνεχίσει να προσφεύγει σε αυτό το σύστημα και να το χρησιμοποιεί μέχρι ότου βρεθεί οριστική λύση μέσα στην επόμενη πενταετία ή τετραετία. Είναι δηλαδή μια προσωρινή λύση αλλά θα πρέπει να βρεθεί κάποια οριστική λύση μέχρι το 2017. Ε, επ' αυτού λοιπόν υπήρξε συμφωνία. Κάποια ειδικά ζητήματα ε, έγιναν αντικείμενο συμφωνίες για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Για αυτές υπάρχει ένας ειδικός εποπτικός μηχανισμός, ούτως ώστε να γνωρίζουμε ποια ευελιξία έχει δοθεί και έχει επιτραπεί σε κάθε λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα και ο ΠΟΕ θα έχει το σύστημα το δικό του για να τις αξιολογήσει και να προτείνει και διαφορετικές ειδικές ε, δυνατότητες ε, ευελιξίας. Έχουμε την παρέκκληση από τις υπηρεσίες στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, δηλαδή το σύστημα επιτρέπει στις πιο πλούσιους χώρες να δίνουν κάποια πλεονεκτήματα στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, ώστε οι τελευταίες να εξάγουν τις υπηρεσίες τους, χωρίς να είναι υποχρεωμένες οι περισσότερο πλούσιες χώρες να δίνουν αυτή τη διευκόλυνση και αυτή τη δυνατότητα και σε άλλες χώρες. Έχουμε κατευθυντήριες γραμμές για την απλούστευση των κανόνων προέλευσης, πολύ τεχνικό ζήτημα, το οποίο όμως κάνει τη διαφορά, ούτως ώστε να μπορέσει μια λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα να εξάγει τελικά στον ε, ε, πιο πλούσιο κόσμο. Τώρα, μίλησε για τη διευκόλυνση του εμπορίου. Η συμφωνία αυτή είναι ένας διεθνής διοικητικός κώδικας για την απλούστευση των τελωνιακών διαδικασιών, για τη έτσι ώστε να γίνει πιο εύκολο να εισάγει κανείς αγαθά σε άλλες χώρες, να μειωθεί η γραφειοκρατία και να αποφευχθούν καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε δυστυχώς εξαιρετικά συχνά. Δηλαδή τα εμπορευματοκιβώτια να είναι κολλημένα για ένα μήνα ε, και στα τελωνία περιμένοντας τη διασάφηση, το, το, το πράσινο φως, ώστε να περάσουν από τα τελωνία. Βεβαίως αυτό ε, είναι πρόβλημα ε, όταν πρόκειται για μηχανολογικό εξοπλισμό που χρειάζονται οι εταιρείε ή όταν πρόκειται για τρόφιμα τα οποία λήγουν. Από εκεί και πέρα Αντιθέτως με το ότι πιστεύετε για τις συμφωνίες του ΠΟΕ, αυτή δεν είναι μια συμφωνία ενός μόνο μεγέθους που θα πρέπει να χωρέσει σε όλους σαν κοστούμι. Είναι πολύ προσεκτικά διατυπωμένη και θα μπορούν να την υλοποιήσουν οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες όποτε μπορούν και κάθε φορά που μπορούν. Άρα οι δεσμεύσεις κατατάσσονται σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες. Μπορείτε να ολοκληρώσετε, διακόπτη πρόεδρος. Ναι, σε ένα δευτερόλεπτο κυρία πρόεδρε. Έχουμε λοιπόν τρεις κατηγορίες συμφωνιών και επιτρέπουμε έτσι στις αναπτυσσόμενες χώρες να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει σε αυτό το πλαίσιο αλλά και να τύχουν στήριξης ώστε να ε, εφαρμόσουν αυτές τις δεσμεύσεις. Δηλαδή έχουμε ένα μέγεθος μεν το οποίο να ταιριάζει σε όλους, αλλά έχουμε και μια εσωτερική διαβάθμιση ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξης ή μη ανάπτυξης της κάθε χώρες οι πιο προηγμένες οικονομίες θα είναι σε θέση να υλοποιήσουν τη συμφωνία σχετικά γρήγορα και αυτό θα ωφελήσει και άλλες αναπτυσσόμενες χώρες και αυτές είναι που θα παρέχουν και την απαραίτητη στήριξη στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Αυτά προς το παρόν για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Θέλετε κύριε Γκάρες το λόγο. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ιδιαίτερα λεπτομεριακή απάντηση που έδωσε και θα μπορούσε να είναι πιο εξονυχιστική αν είχαμε περισσότερο χρόνο. Μήπως θα μπορούσατε να μας δώσετε και γραπτό στην απάντησή σας, γιατί νομίζω ότι ενδιαφέρει όλα τα μέλη της Επιτροπής μας. Και μας ενδιαφέρουν όλες οι λεπτομέρειες ε, που δώσατε κυρίως ε, στο τελευταίο τμήμα για τις τρεις διαφορετικές κατηγορίες δεσμεύσεων που αναλάβαμε στον Παλί. Όλους μας ενδιαφέρει το θέμα και θέλουμε να είμαστε ενημεροί. Ευχαριστώ. Ωραία. Θα ήθελα να καλωσορίσω τώρα το Γενικό Διευθυντή τη Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ, τη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστική Βοήθεια, τον κύριο Κλάου Σόρενσεν, που θα μα ενημερώσει για την κατάσταση μετά την επιδείνωση της κρίσης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και τη Συρία. Δυστυχώς ε, δημιουργήθηκε μια νέα διάσταση της κρίσης ε, που χρήζει της άμεσης ε, προσοχής μας. Το Δεκέμβριο στο Νότιο Σουδάν οι πολιτικές εντάσεις ε, κλιμακώθηκαν, είχαμε βιοπραγίες και μια δυστυχώς μεγάλη επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης. Πάνω από 400.000 άτομα εκτοπίστηκαν και είχαμε χιλιάδες ε, νεκρούς και τραυματίες. Ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Σόρενσεν για 20 λεπτά. Λυπούμε, αλλά δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κυρία Ζανίκη και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να ενημερώσω την Επιτροπή σας για τρεις ε, εξαιρετικά σοβαρές ανθρωπιστικές κρίσεις που εκτιλήσονται την ώρα που μιλάμε. Νομίζω ότι το όλο σύστημα πασχί, πασχίσει να αντιμετωπίσει αυτές τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Έχουμε μια ασυνήθιστη κατάσταση με τρεις κρίσεις ε, εκτάκτου ανάγκης επίπεδου 3 όπως έχει κρίνει και ο ΙΕ και οι, οι διάφορες οργανώσεις. Έχουμε την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, τις Φιλιππίνες και τη Συρία. Και επιπλέον έχουμε και τα γεγονότα στο Νότιο Σουδάν που προστίθενται στις τρεις προηγούμενες κρίσεις που έχουν φέρει τα πάνω κάτω ουσιαστικά. Και είναι πολύ δύσκολο και περίπλοκο να αντιμετωπίσουμε ταυτόχρονα όλες αυτές τις ε, δρυμύτατες ανθρωπιστικές κρίσεις. Σας διαβεβαίω πάντως ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε, βάζουμε τα δυνατά μας και θα ήθελα να πω ότι όλες οι προσπάθειες που κάναμε προκειμένου να μετατρέψουμε και να δρομολογήσουμε τις ε, ανθρωπιστικές επιχειρήσεις ε, των φορέων του ΟΗΕ σε αυτή την μεταβατική ατζέντα αρχίζει και αποδίδει καρπούς η νέα προσπάθεια. Και το νέο εργαλείο με, την, με το χαρακτηρισμό της κρίσης επίπεδου 3 και η άμεση κινητοποίηση προσωπικού από άλλες, από άλλες λιγότερο οξύες καταστάσεις και η στελέχωση με πολύ δυναμικούς ανθρώπους, όχι μόνο από την Ότσα, αλλά και από όλους τους οργανισμούς και τις υπηρεσίες του ΟΗΕ, όλες αυτές οι προσπάθειες αρχίζουν και αποδίδουν. Έχουμε λοιπόν αλλαγές που μας δίνουν έστω και μικρές ελπίδε για το μέλλον. Θα ήθελα επίσης να πατήσω φόρο τιμή στους συνεργάτες μου, γιατί στο Νότιο Σουδάν κάποιοι εταίροι μας στον ανθρωπιστικό τομέα απέστειλαν το προσωπικό τους. Εμείς παραμείναμε εκεί. Κρατηθήκαμε και ήταν πολύ σημαντικό για μας να έχουμε μέσα των συνεργατών μας μάτια και αυτιά επιτόπου στη, στο Νότιο Σουδάν, ώστε να συνεχίσουμε τις επαφές με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, να κρατήσουμε ακμαίο το ηθικό του τοπικού πληθυσμού και να μην ξεφύγουμε από το στόχο μας. Η κατάσταση δεν ήταν καθόλου εύκολη και μάλιστα θα πρέπει να δώσω άδεια στους μερικούς συνεργάτες μου, ιδιαίτερα όσοι επέστρεψαν από την Τζούμπα που η κατάσταση ήταν πραγματικά δερημήτατη. Πάντως αλλάζουμε συνέχεια το προσωπικό, απομακρύνουμε μερικούς, ε, πούμε άλλους, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις θα ήθελα και σε αυτές να πω ότι φόρο τιμή, γιατί κρατιώνται εκεί με νύχια και με δόντια. Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα συγκεκριμένα, γιατί είναι πάρα πολλέ οι μη κυβερνητικέ οργανώσει. Πραγματικά χρειάζεται μεγάλο θάρρο για να μείνει κανεί ε, στο Νότιο Σουδάν, ιδιαίτερα σε απομονωμένε περιοχέ, γιατί ε, κανείς δεν ξέρει αν πάνε στραβά τα πράγματα, αν θα τους α, α, μπορέσει να τους απομακρύνει κανένας, αν θα μπορούν να κατεβούν, να προσγειωθούν ελικόπτερα και να τους βοηθήσουν να επιστρέψουν. Και μάλιστα Ακριβώ επειδή είχαμε κάποιε αερογέφυρε ανθρωπιστική βοήθεια, δείξαμε τη στρατηγική μα αξία. Σε μερικέ περιπτώσει που είχαν ακυρωθεί όλε οι πτήσει και είχαμε ελάχιστε δυνατότητε αερομεταφορά, εμεί καταφέραμε να προσγειώσουμε εκεί αεροπλάνα και να κατορθώσουμε να φτάσει εκεί η ανθρωπιστική μας βοήθεια, το προσωπικό, ε, υπάλληλοι ανθρωπιστικών φορέων και να βοηθήσουμε να απομακρυνθούν άλλοι που έπρεπε να φύγουν. Δημιουργήθηκε λοιπόν ένα δίκτυο ασφαλείας ε, εκεί που ήταν πολύ χρήσιμο για όλους τους εργαζόμενους εκεί. Τώρα με δύο λόγια θα ήθελα να πω μερικά πράγματα για τις τρεις διαφορετικές ε, κρίσεις. Για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία ειλικρινά ήταν αναμενόμενα τα πράγματα εκεί. Και ίσως ε, ένα παράπονο που θα είχα να κάνω ήταν ότι το σύστημα δεν έλαβε δεόντως υπόψη και έγκαιρα τα, τους διάφορους συναγερμούς ώστε να κινητοποιήσουμε σταθεροποιητικούς μηχανισμούς το συντομότερο δυνατό. Ήταν κάτι που το βλέπαμε να έρχεται, αλλά αυτό θα πρέπει να μας γίνει μάθημα για το μέλλον, γιατί κάτι παρόμοιο είχαμε σχεδόν και στο Μαλί και στο Νότιο Σουδάν ε, μας κατέλαβαν εξαπίνης μερικές φορές. Στον Μπάνγκουι όμως και στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία παρακολουθήσαμε τα πράγματα σε πραγματικό χρόνο. Βλέπαμε τις ειδήσεις τηλεόραση, οπότε ξέρετε την κατάσταση, δεν έχω να σας πω και πολλά. Πάντως αυτό που προκύπτει από την ανάλυση είναι ότι η αιτία της κρίσης δεν είναι θρησκευτική. Είναι η μαζική επανάπτυξη είναι ότι οι άνθρωποι δεν έχουν μέσα βιοπορισμού, δεν ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν το μέλλον τους και προσβλέπουν προς την κυβέρνηση, προς τον Μπαγκουή, την πρωτεύουσα για βοήθεια, αλλά βοήθεια δεν φτάνει. Γι' αυτό και ξεκίνησαν οι εξεγέρσεις, ε, οι ανταρσίες και όταν έχουμε μαζική ανεργία κυρίως των νέων και είδατε ε, οι άνθρωποι παίρνουν τα δρεπάνια και τα ματσέτες, ε, δημιουργείται μια κατάσταση και οι προϋποθέσεις για τον όλεθρο. Και δυστυχώς αυτή η κατάσταση δημιουργεί μια παλινδρόμηση στις εθνοτικές και τις ε, θρησκευτικές ρίζες. Γι' αυτό και είναι τόσο επικίνδυνη η κατάσταση. Κάτι που οφείλεται σε τελική ανάλυση στην επανάπτυξη μετατρέπεται σε μια σύγκρουση θρησκειών, θρησκευμάτων ή ε, σε σύγκρουση που έχει εθνοτικές ε, ρίζες. Ο συνολικός αριθμός των εκτοπισμένων, όπως μας είπατε κυρία Πρόεδρε, είναι γύρω στις 25 με 30% του συνολικού πληθυσμού. Φανταστείτε τι θα αντιπροσώπευε ένας τέτοιος αριθμός στο Βέλγιο. Δύο εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισθέντων ανθρώπων που διακινούνται μέσα στο Βέλγιο και δεν ξέρουν πού να πάνε. Και η κατάσταση δεν βελτιώνεται. Έχουμε μια εξαιρετικά ρευστή κατάσταση στους καταβλισμούς ε, των προσφύγων και μιλάμε πολλές φορές ε, στη Δύση για την κατάσταση στα αεροδρόμια και το λέμε γιατί εκεί δημιουργούνται δυσκολίες στην άφηξη της ανθρωπιστικής βοήθειας και στην άφηξη των, ε, ανθρωπιστικών οργανώσεων. Πρέπει να περάσουν από το αεροδρόμιο του Μπάγκου και αν έχουμε 100-120 ε, εσωτερικά εκτοπισμένους που κατασκηνώνουν στην περιοχή του αεροδρομίου δεν μπορούν να προσγειωθούν τα αεροπλάνα. Γι' αυτό και είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να επισημάνω, γιατί θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τη στέγη της Κινές, τα, τα, τα ζητήματα προστασίας, την παροχή υδατος. Τώρα οι μουσουλμάνοι βρίσκονται στο στόχαστρο, κακοποιούνται, τους βγάζουν από τα φορτηγά, τους κατεβάζουν, δεν μπορούν να προχωρήσουν αλλά ε, επίσης έχουν ε, καταστραφεί τα αποθέματα σπόρων. Έχουν καεί. Οπότε περιμένουν την επόμενη συγκομιδή ε, που και αυτή διατρέχει κίνδυνο. Έχουμε πολλές προτεραιότητες, θα πρέπει να τις ιεραρχήσουμε. Πάντως, μία από τις σημαντικές προτεραιότητες είναι να φτάσουν σπόροι στη χώρα ώστε να εξασφαλιστεί, να εξασφαλιστεί ένας ελάχιστος βαθμός ασφάλειας για να μπορούν οι γεωργοί να φυτέψουν τους σπόρους αυτούς. Αλλιώς θα έχουμε μετά από ένα εξάμεινο, μετά την περίοδο των βροχών και το καλοκαίρι, θα έχουμε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση και θα πρέπει να αντισταθμίσουμε με μαζικές παροχές επισητιστικής βοήθειας. Και μια και σπανίζουν οικονομικοί πόροι, γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς που έχουμε προβλήματα και άλλοι δωρητές έχουν πρόβλημα. Θα πρέπει να αποφύγουμε λοιπόν με έγκαιρη πρόληψη για τις σπορές ε, την κατάσταση αυτή. Κάτι άλλο που θα πρέπει να έχουμε υπόψη είναι η απόλυτη ανάγκη ασφάλειας. Βρέθηκα σε μια παράδοξη κατάσταση προχθές ε, όταν ενημέρωσα τον αρμόδιο επίτροπο στο Συμβούλιο και είπα ότι ε, δεν θα περιμένατε ένα τέτοιο σχόλιο από μένα γιατί εργάζομαι στον ανθρωπιστικό κλάδο, αλλά οι μη κυβερνητικέ οργανώσει σα οικετεύουν να εξασφαλίσετε τέτοια ασφάλεια. Ουσιαστικά ζητούν μια ισχυρότερη στρατιωτική παρουσία για να αποκατασταθεί ασφάλεια. Δεν θέλουν γιατί θέλουν να στηριχθούν στο στρατό, αλλά χωρί στοιχειώδη ασφάλεια δεν μπορούν ότι οι ανθρωπιστικέ οργανώσει να παραδώσουν την επισητιστική βοήθεια, φάρμακα, νερό. Και η ρευστή κατάσταση στη χώρα είναι τόσο προφανής ώστε χρειάζεται μια τέτοια σταθεροποίηση με τη βοήθεια ίσως του στρατού. Δεν είμαι ευτυχής που λέω κάτι τέτοιο, αλλά παρηγοριάμαι από δύο τινά. Καταρχήν πιστεύω ότι σήμερα στο Συμβούλιο θα η απόφαση για την αποστολή της ΚΕΠΑ, ούτε και αυτή ήταν ε, βέβαιη, γιατί έγιναν πολλές συζητήσεις και στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο και για τις ε, ομάδες μάχης Ελπίζω όμως, ευελπιστώ, ότι στα συμπεράσματα του Συμβουλίου θα ληφθεί και τέτοια απόφαση. Και επίση θα ανακύψει το ερώτημα ποιο θα το αναλάβει κάτι τέτοιο. Πάντως το μήνυμα ότι χρειαζόμαστε ασφάλεια νομίζω ότι έχει γίνει αντιληπτό από όλους και θεωρώ ότι θα γίνει κάτι. Οι Γάλλοι αναλαμβάνουν ένα τεράστιο βάρο στην όλη κατάσταση θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε, αλλά και οι Αμερικανικά εξασφαλίζουν κάποιες αερογέφυρες για να βοηθήσουν τα αφρικανικά στρατεύματα να διακινηθούν. Πάντως ε, θα πρέπει να αναλυθεί δράση το συντομότερο δυνατό για την ασφάλεια. Ένα άλλο βραχυπρόθεσμο ζήτημα είναι και ο αφοπλισμός, γιατί από τη στιγμή που έχουμε νέους που μετακινούνται με διάφορα όπλα και ο στρατός δεν θα βρίσκεται παντού η στρατιωτική παρουσία δεν θα εξασφαλιστεί παντού. Οπότε θα δημιουργηθεί πολύ σοβαρός κίνδυνο για τον άμαχο πληθυσμό. Αυτό ίσως θα ήταν το δεύτερο σημείο και δεν ε, αφορά αμυγό την ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά είναι προϋπόθεση για την ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει στον προορισμό της, η ασφάλεια. Κάτι άλλο που θα πρέπει να έχουμε υπόψη, και αυτό φυσικά ξεφεύγει από τα ανθρωπιστικά, αλλά κάποιο θα πρέπει να το σκεφτεί. Πώ θα εξασφαλιστεί ε, η επιβίωση των ε, στρατιωτών και αν έχουμε 2.000 στρατιώτες νηστικούς, τότε διάφοροι άλλοι κίνδυνοι και απειλές ε, θα ανακύψουν. Θα πρέπει και αυτό να το λάβουμε υπόψη λοιπόν. Επίσης, ε, θα πρέπει να ξαναλειτουργήσουν οι ραδιοφωνικοί σταθμοί. Να φτάσει το μήνυμα προς τα χωριά, προς το πληθυσμό για να καταλάβει ο κόσμος ε, τι συμβαίνει. Τα καλά μαντάτα είναι ότι έχει ξεκινήσει μια πολιτική διαδικασία και ευελπιστώ θα ότι θα επιβεβαιωθεί και από τον Πρόεδρο να δοθεί μια προοπτική. Ακόμη και αν είναι χαλαρή, να δοθεί μια προοπτική ότι κινούμαστε προς τις εκλογές για να ξαναρχίσει η ανοικοδόμηση, η ανασυγκρότηση της χώρας. Και τα λέω όλα αυτά γιατί οι φορείς των ανθρωπιστικών οργανώσεων δεν μπορούν να επιτελέσουν το έργο τους σε μια χαοτική κατάσταση. Όσο κουράγιο να έχουν και να πηγαίνουν στα χωριά, όταν φεύγουν από τα χωριά, όταν εγκαταλείπουν το χωριό, η κατάσταση καταραίει. Ε, ένα άλλο καλό νέο και ε, γύρισα από μια ομάδα υψηλού επίπεδου, γι' αυτό και δεν ήρθε εδώ κυρία Γεωργίευα. Πηγαίνει από συνεδρία σε συνεδρίαση για να συμπεριληφθεί η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία στα συμπεράσματα του Συμβουλίου και μετά θα έρθει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να σας εξηγήσει την κατάσταση. Τα καλά νέα πάντως είναι ότι υπήρξε προθυμία και βούληση να δοθεί υπόσχεση για 500 εκατομμύρια, μισό δισεκατομμύριο δολάρια. Θα είναι γύρω στα 400 εκατομμύρια δολάρια υπόσχεση δωρεάς που θα είναι ένα συνδυασμό αναπτυξιακών κονδυλίων και κονδυλίων για ανθρωπιστική βοήθεια. Και ένα τμήμα τους είναι δωρεά ένα μικρό τμήμα θα έχει τη μορφή μακροπρόθεσμων δανείων από την Παγκόσμια Τράπεζα. Πάντως ε, θα είναι αρκετά γενναιόδορη ανάληψη υποχρέωση ε, δέσμευση τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να βελτιώσει την κατάσταση εκεί και με ευφύ τρόπο. ό,τι αφορά το συντονισμό ε, τη ανθρωπιστική βοήθεια, και αυτό έχει ξεκινήσει. Έχουμε εξασφαλίσει ηγετικό ρόλο εκεί, χαίρομαι. Έχουμε οργανώσει καλά τα πράγματα και άκουσα ότι υπάρχει δυνατότητα για μία αναβάθμιση, οπότε τα επιπλέον κονδύλια που προτείνονται θα δοθούν για αναβάθμιση του συντονισμού και της οργάνωσης σε διάφορα σημεία. Το μείζον πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε αρκετή παρουσία στις διάφορες επαρχίες και εκεί είναι που υπάρχει πιο οξύ πρόβλημα ασφάλειας αν απομακρυνθεί κανείς 100 με 200 χιλιόμετρα από τον Μπάγκου ή την πρωτεύουσα, τότε βλέπουμε ότι η κατάσταση είναι αρκετά επισφαλής. Αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε. Μισό δισεκατομμύριο δολάρια, δηλαδή 500 εκατομμύρια δολάρια, αποστολή και ΠΑ, προθυμία για ανάληψη δράσης. Πιστεύω ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση και επίσης θα πρέπει να σταθεροποιήσουμε ή να να δημιουργηθεί μια νέα κυβέρνηση γιατί έχουν καταστραφεί τα αρχεία, έχουν εξαφανιστεί, ε, λαιλατηθεί ε, τα αρχεία, έχουν εξαφανιστεί υπουργοί. Υπάρχει ένα κενό. Θα πρέπει να διδαχθούμε από τα μαθήματα του Μαλί και της ε, Σομαλίας. Δεν ξέρω, κάποια, κάποιες συμβάσεις για την ανασυγκρότηση των υποδομών, κάποια στοιχεία από εκεί να τα αξιοποιήσουμε και εδώ για να δώσουμε σε αυτό το φτωχό κόσμο νέες προοπτικές. Τώρα, Νότιο Σουδάν. Προφανώς, σας φαίνεται κάπως παράξενο και εμένα μου φαίνεται παράξενο το ότι δεν αποκλήθηκε η κρίση αυτή, η κρίση επίπεδου 3, παρόλο που τα χαρακτηριστικά της προσυδειάζουν σε μια κρίση επίπεδου 3. Δεν είμαι σίγουρος ότι καταλαβαίνω ακριβώς το γιατί και θα ρωτήσω και θα επανέλθω. Από όσο γνωρίζω, δεν τη λέμε κρίση επίπεδου 3, γιατί προϋπήρχε πριν και ε, απέκτησε τεράστιες διαστάσεις. Γι' αυτό δεν αποκτά αυτό το όνομα το επίσημο, αν θέλετε. Έχουμε τον Τόμπι Λάνσεν, συντονιστή για θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας. Έμεινε ακόμα και όταν το UNTSS ζητούσε από όλους να εγκαταλείψουν τη χώρα, Έμεινε λοιπόν και ήδη όλη την κρίση και η δική μου μιας άνθρωποι παρέμειναν παρόλο που οι πυροβολισμοί ε, έπεφταν προ βροχή. Και ελπίζουμε ότι οι συζητήσεις στην Άντις θα ε, πετύχουν, θα καταλήξουν σε μια κάποια ε, πρόοδο. Θέλω να ευχαριστήσω τον Άλεξ Ρόντο, ειδικό απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιτόπου, ο οποίος εξασφαλίζει ε, ότι το περιεχόμενο της Ειρηνευτικής Συμφωνίας ή εν πάση της Συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός θα συνάδει με τους βασικούς κανόνες για τα θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας. Ε, δεν είναι εύκολο, αλλά τα παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς, όσο περισσότερο μπορούμε. Δεν έχουμε ακόμα επιταχύνει την χρηματοδότησή μας, διότι ήδη είχαμε αναλάβει πολύ μεγάλη οικονομική δέσμευση στο Νότιο Σουδάν. Τι κάνουμε, αναθεωρούμε, επανεξετάζουμε τις ε, αξιολογήσεις που έχουμε για τις διάφορες ανάγκες που υπάρχουν για να καταλάβουμε πού πρέπει να δώσουμε βάρος αν τελικά επιβεβαιωθεί ότι κάτι πρέπει να γίνει. Θα ήθελα λοιπόν σε αυτό το σημείο να σας εφιστήσω την προσοχή σε μια πολύ μεγάλη ανησυχία που είναι μας χαρακτηρίζει αν θέλετε, από τη στιγμή που είναι μαζική η ανασφάλεια στο νότιο Σουδάν, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για όσους εργάζονται στον τομέα της ανθρωπιστικής βοηθείας να τοποθετήσουν εκ των προτέρων ε, τα τρόφιμα και τα φάρμακα πριν την περίοδο των βροχών. Θα είναι δύσκολο λοιπόν να τα διανύμουν και αν δεν γίνει αυτό τότε η κατάσταση θα δυσκολέψει πάρα πολύ. Γιατί μετά όταν θα ξεκινήσει η περίοδος των βροχών μόνο με ελικόπτερο μπορεί να μεταφερθεί ε, το οποιοδήποτε τρόφιμο και αυτό είναι απαγορευτικά ακριβό. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε σταθεροποίηση τώρα, πριν την περίοδο των βροχών. Πρέπει να συμφωνήσουν σε κατάπαυση πυρός τώρα και είναι η μόνη προϋπόθεση ούτω ώστε να ε, μεταφέρει και να δρομολογήσει τα διάφορα αποθέματα ΟΗΕ στις διάφορες ε, περιοχές της χώρας. Βέβαια έχουμε μαζικές καταστρατηγήσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων, ελοχεύει ο κίνδυνος σύγκρουσης μεταξύ των ΝΟΥΡ και των ΠΙΝΚΑ, ε, έχουμε εθνοτικές ομάδες με πολύ περίπλοκες σχέσεις μεταξύ τους. Αυτά για το Νότιο Σουδάν, για τη Συρία. Νομίζω ότι παρακολουθήσατε όλη τη διάσκεψη των δωρητών στο Κουβέιτ και που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα και στο, το Σαββατοκύριακο γνωρίζουμε ε, τι συνέβη με τη συμμετοχή της αντιπολίτευσης στη Γενέβη 2, ε, μια διάσκεψη που θα ξεκινήσει ο Σονούπο. Καλό νέο αυτό. Άλλο καλό νέο είναι ότι τουλάχιστον μέρος της αντιπολίτευσης επιθυμεί να συνεργαστεί. Δύο λεπτά ακόμα χρειάζομαι κυρία Πρόεδρε. Και τρίτο καλό νέο είναι ότι η διάσκεψη στο Κουβέιτ κατέληξε σε μαζική ανάληψη δεσμεύσεων για τη συνέχιση της χρηματοδότησης ε, στη χώρα αυτή. Δεν είναι εύκολο, σίγουρα. Όλοι ελπίζουμε ότι θα δούμε το φως στην άκρη του τούνελ μετά τη Γενέβη 2. Όλοι έχουμε αμφιβολίες και καλώς. Σαφέστατα όμως, όλοι όσοι εργαζόμαστε στον ανθρωπιστικό ε, κλάδο αναρωτιόμαστε πότε θα πρέπει να ανέβουν οι τόνοι στη ρητορική εν πάση περιπτώσει. Διότι ο όγκος των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρωπιστικής νομοθεσίας είναι τεράστιος. Ασχολούμαστε λοιπόν με το φάκελο της Συρίας. Ε, ε, συστήσαμε την ομάδα υψηλού επίπεδου για την πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια. Κάποια μικρά αποτελέσματα έχουν αρχίσει να έρχονται, αλλά σταματήσω κάπου εδώ. Ναι, θα σας δώσω λίγα λεπτά ακόμα αν θέλετε, λέει η πρόεδρος μάλιστα. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να σας δώσω και άλλα 20 λεπτά, αλλά ο χρόνος μας πιέζει και έτσι δυστυχώς ε, δεν μπορώ να σας δώσω παραπάνω χρόνο. Ο κύριος Γκέρενς για ένα λεπτό μόνο παρακαλώ. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Γκέρενς. Έχω μία ερώτηση για το θέμα της χρηματοδότησης. Ο κύριος Σέρενσεν είπε ότι καλά είναι τα νέα και θα πρέπει να χαρούμε. Την περασμένη εβδομάδα ε, όμως ο κόσμος των ανθρωπιστικών οργανώσεων μας είπε ότι τα χρήματα δεν θα έφταναν και ότι θα πρέπει να δώσει απάντηση η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μίξη, τη μεικτή χρήση ε, κονδυλίων από το, την ανάπτυξη και κονδυλίων από την ανθρωπιστική βοήθεια ε, στο θέμα του Μπαγκή. Ε, σας ερωτώ, τα κονδύλια που χρηματοδοτούν όλες αυτές τις δράσεις στο βαθμό που ανήκουν στο Ταμείο για την Ανάπτυξη εξυπηρετούν αυτό το σκοπό της ανάπτυξης ή μήπω είναι ένα μέτρο έτσι ώστε να παίρνουμε το Ταμείο της Ανάπτυξης τα χρήματα που μας λείπουν από το Ταμείο της Ανθρωπιστικής Βοήθειας. Δεν ξέρω αν με καταλάβατε και δεύτερον, δεύτερο ερώτημά μου είναι το εξής. Σε ποιο βαθμό ε, η διευκόλυνση αυτή και τα εργαλεία που έχουν δοθεί στην Αφρικανική Ένωση αξιοποιούνται για να έχουμε χρηματοδότηση στρατιωτικών δράσεων. Γίνεται κάτι τέτοιο στον Ταρφούρ. Γνωρίζουμε ότι αυτό το ταμείο χρησιμοποιήθηκε για να συμβάλλει ούτως ώστε η Αφρικανική Ένωση να αναλάβει τις στρατιωτικές της υποχρεώσεις στην περιοχή. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φυσικά δεν προλαβαίνω σε δύο λεπτά να αναλύσω όλο αυτό το πρόβλημα, αλλά ευχαριστώ για την ενημέρωση. Ακούσαμε Πολλέ πληροφορίε για πολλά τα δεν αναφερθήκατε αρκετά στον ανθρώπινο παράγοντα. Μιλήσατε για την ελπίδα. Δύο φορέ αναφέρατε την ελπίδα. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Και είπατε και κάτι άλλο σημαντικό. Το, το πρόβλημα δεν είναι θρησκευτικό. Το πρόβλημα είναι πρόβλημα υπανάπτυξη. Και πραγματικά εκεί θέσατε το δάκτυλο επί των τύπων των ήλων. Ε, θα πρέπει να γίνει καλός έλεγχος αυτών των κονδυλίων. Επίσης είπατε ότι ευχαριστείτε και τη Γαλλία και τη θέση στο Μαλί. Ξέρετε όμως ότι τι γίνεται όταν αποσύρεται ο στρατό. Τι γίνεται στο βόρειο Μάλι που έχει αποχωρήσει ο στρατό. Επανέρχονται οι συμμορίε και μάλιστα ετοιμάζονται να πάνε και στη Λιβύη. Οπότε δεν ε, ετοιμάσαμε τη μετάβαση μετά την αποχώρηση του στρατού. Τι γίνεται. Εκεί είναι το πρόβλημα στο Μάλι. Επίση, μιλήσατε για την ανασυγκρότηση των κρατικών θεσμών και δομών. Και στο Νότιο Σουδάν έχουμε και το πρόβλημα του Σαχέλ. Ε, είναι χώρες ε, και το Νότιο Σουδάν που έχει πολύ πλούσιο ρηκτό πλούτο. Το υπέδαφος είναι πολύ πλούσιο, αλλά δυστυχώς ε, ο πλούτος αυτός δεν ωφελεί τον τοπικό πληθυσμό. Το υπέδαφος είναι πάμπλουτο και η χώρα είναι πάμφτωχη. Ο κόσμος είναι φτωχός. Πιστεύω πάντως ότι αξίζεται συγχαρητηρίων γιατί για μία ακόμη φορά, για μία φορά είπατε την αλήθεια, δεν εννοώ εσάς προσωπικά, αλλά πραγματικά ε, είπατε τα πράγματα με το όνομά τους. Και όταν βλέπουμε τον Νότιο Σουδά βλέπουμε ότι δεν είναι και τόσο μακριά από την Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ ρεαλιστές και να περιγράφουμε με ρεαλισμό τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Κύριο Σόρενσεν. Έχετε ένα-δύο λεπτά για τις απαντήσεις. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Δεν πρόκειται εδώ τώρα να μεταφέρουμε κονδύλια από, το, από την ανάπτυξη στον ανθρωπιστικό κλάδο. Γιατί αυτό φοβάστε. Δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο, σας ε, διαβεβαιώ. Τώρα, τι συνέβη στο Μαλί. Μια και οι διαδικασίε στην ΔΕΦΚΟ μερικέ φορέ είναι πιο χρονοβόρε. εγώ δέχτηκα να αναλάβω ένα ε, μικρό κονδύλιο για να ε, ξεκινήσουν και πάλι τα σχολεία. Έχουμε διάσταση και αναπτυξιακή. Γιατί ε, για, την, για τους μισθούς, για τα σχολεία, κάναμε κάτι που βρίσκεται στο περιθώριο ουσιαστικά της ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά το κάναμε για να βοηθήσουμε έχει έντονο αναπτυξιακό χαρακτήρα και το θέμα της ε, προσαρμοστικότητας, της ανθεκτικότητας, ε, Εκεί είναι συναφής οι δύο κλάδοι της ανάπτυξης και της ε, ανθρωπιστικής βοήθειας. Γιατί αν η ανάπτυξη δεν ξεκινήσει, θα είναι πολύ πιο έντονο το βάρος για την ανθρωπιστική βοήθεια. Αν μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους αρμόδιους για την ανάπτυξη να ξανακοινοτοποιήσουν την οικονομία, όλα καλά. Γι' αυτό και ο Άντριος Πίπερ και η Κρυσταλίνα Γεώργιεβα συνεργάζονται στενά. Σε ό,τι αφορά τις διευκολίες και τα εργαλεία για την ειρήνη, δεν έχω στοιχεία, δεν γνωρίζω την αλήθεια. Αν κάποιος άλλος τη γνωρίζει, ε, να σας ενημερώσει. Εγώ δεν έχω εδώ πρόβλημα. Θα ενημερωθώ και θα σας τη στείλω γραπτός. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει μία αμυγός ανθρωπιστική απάντηση. Η απόκριση, η αντίδραση θα πρέπει να είναι εκείνη, αναπτυξιακή και ανθρωπιστική. Στην κεντροαφρικανική δημοκρατία θα καταφέρουμε μέσω μία στοιχειώδη πολιτική ασφάλεια να εξασφαλίσουμε στοιχειώδεις ε, κρατικούς θεσμούς. Θα πρέπει και οι δύο πυλώνες, και οι δύο βραχίονες, και ο αναπτυξιακός και ο ανθρωπιστικός να συνεργαστούν. Κύριε Γουατά, Νομίζω ότι έτσι απάντησα και στη δική σας ερώτηση. Χωρίς ανάπτυξη θα έχουμε τέτοια προβλήματα. Η πανάπτυξη είναι η αιτία που ενισχύεται από την έλλειψη ασφάλειας. Αναφέρατε τη Λιβύη, τη συνέβη στη Λιβύη. Εκεί πραγματικά είχαμε ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Και σε τελική ανάλυση μας ενδιαφέρει η ανάπτυξη, η αποκατάσταση της ανάπτυξης. Και θα πρέπει να γίνει σχετική συζήτηση, γιατί η χρηστή διακυβέρνηση βρίσκεται στο επίκεντρο της κατάστασης, γιατί με ε, μια σωστή χρηστή διακυβέρνηση, με ένα σύστημα πιο περιεκτικό που δεν θα αποκλεί κανέναν και με τον πληθυσμό που θα είναι αποδέκτης ενός τμήματος τουλάχιστον ε, του πλούτου των πόρων, θα βελτιώσουμε την κατάσταση. Αν συγκρίνουμε τις ε, επενδύσεις και τα άλλα κονδύλια, η αναπτυξιακή βοήθεια είναι ένα μικρό κλάσμα όλων αυτών. Αλλά χρειάζονται όλα αυτά θα πρέπει να είμαστε πιο εστιασμένοι στις αναπτυξιακές δράσεις όπως το κάνουμε και στις ανθρωπιστικές. Και είμαι στη διάθεσή σας για τη συνέχεια της συζήτησης που είναι πραγματικά συναρπαστική γιατί η κατάσταση όντως είναι επικίνδυνη για την Ευρώπη. Σας ευχαριστούμε εκ βάθους καρδίας κύριε Σόρενσεν γιατί πραγματικά η παρέμβασή σας ήταν καταπληκτική. Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο για τη συζήτηση, δυστυχώς ε, έχει εξαντληθεί και ζητώ συγγνώμη και από τον κύριο Λάστρα γιατί θα χρειαστεί να αναβάλουμε για αύριο την ε, έκθεσή του με θέμα την εξάλληψη των βασανιστήριων στον κόσμο. Σας ζητώ συγγνώμη κύριε Λάστρα, αλλά έχουμε εξαντλήσει το χρόνο για τα υπόλοιπα θέματα. Θα επανέλθουμε στην έκθεσή σας ε, αύριο το πρωί. Θα είναι το πρώτο θέμα αμέσως μετά τη συνεδρίαση των συντονιστών. Λυπούμε, αλλά ο χρόνος ε, μας πιέζει. Και πρέπει να σε αφήσω γιατί θα πρέπει να πάω στο Παρίσι. Αύριο θα έχουμε και τις ψηφοφορίες. Θα τα ξαναπούμε αύριο.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 Euh, Κυρίες και κύριοι, θα ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της ε, απογευματινής μας συνεδρίασης. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Χαίρομαι διότι σας καλωσορίζω σήμερα στην ακρόαση με αντικείμενο τη θέση της ανθρωπιστικής βοήθειας στην εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η σημασία του σεβασμού των ανθρωπιστικών αρχών. Χαίρομαι επίσης όλους τους παρεμβε... ε, διότι έχουμε όλους παρεμβαίνοντες ε, εδώ και τους ευχαριστώ θερμά. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Δεκέμβριο του 2013 παρουσίασαν μια ανακοίνωση για τη συνολική προσέγγιση που θα πρέπει να ακολουθείτε ε, σε αυτές τις συγκρούσεις και θα πρέπει να είναι στρατηγικός συνεκτική η προσέγγιση με συνεκτικό τρόπο να χρησιμοποιούνται τα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ένωση έχει πάρα πολλές πολιτικές, εργαλεία, μέσα και δράσεις από τη διπλωματία μέχρι την ανθρωπιστική βοήθεια διαμέσου της ασφάλειας, της άμυνας, της χρηματοδότησης, του εμπορίου και της συνεργασίας για την ανάπτυξη. Έχει λοιπόν όλα αυτά τα μέσα στη διάθεσή της. Είναι η πρώτη εμπορική δύναμη στον κόσμο, η Ευρωπαϊκή Ένωση και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 είναι και ο μεγαλύτερος δωρητής για θέματα ανάπτυξης και για ανθρωπιστική βοήθεια. Η συνθήκη της Λισαβόνας ε, κατοχυρώνει την ιδιαιτερότητα της ανθρωπιστικής ε, βοήθειας και ανθρωπιστικής δράσης. Ε, απαιτούνται οι αρχές της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας. Η τήρηση και ο σεβασμός αυτών των αρχών είναι απαραίτητα για να είναι αποτελεσματική η ανθρωπιστική δράση και για να είναι ασφαλής όσοι ασχολούνται με αυτή. Διότι το να υπάρχει σχέση μεταξύ πολιτικών στρατιωτικών στόχων και της ανθρωπιστικής βοήθειας μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τους λειτουργούς της ανθρωπιστικής βοήθειας. Η ιδιαιτερότητα λοιπόν της ανθρωπιστικής βοήθειας είναι προφανής και τονίζεται στην ανακοίνωση. Με τη σημερινή ακρόαση θα ε, διερευνήσουμε τη θέση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη συνολική προσέγγιση. Θα μιλήσουμε για τα διδάγματα που έχουμε αντλήσει επί τόπου. Να δώσω καταρχάς τον λόγο στον κύριο Νόρμπερτ Νόιζερ, ο οποίος θα προεδρεύσει σε αυτή την ακρόαση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε και κύριοι. Και εγώ θα ήθελα να σας καλωσορίσω με τη σειρά μου στην ακρόαση που θα έχουμε σήμερα. Θα έχουμε δύο πάνελ. στο πρώτο πάνελ θα ασχοληθούμε με ένα γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο ασκούν τα καθήκοντά τους η λειτουργή της ανθρωπιστικής βοήθειας και στο δεύτερο πάνελ θα ασχοληθούμε με πιο συγκεκριμένες περιπτώσεις και θα προσπαθήσουμε να αντλήσουμε κάποια διδάγματα για το μέλλον. Ελπίζω λοιπόν να είναι πολύ επικοδομητική η ακρόση για όλους σας. Πρώτος ε, ομιλητής θα είναι ο κύριος Κλάους Σόρενσεν, Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης για την Ανθρωπιστική Βοήθεια. Έχετε το λόγο κύριε Σόρενσεν για 7 λεπτά. Εδώ είμαι. Αλλά... Αλλού σας έψαχνα. Ε, συνέχεια κινούμε. Έτσι έχω προγραμματιστεί και γενετής. Ίσως αυτή τη φορά σε αυτήν την ομιλία δεν χρειάζεται καν να εξαντλήσω το χρόνο που μου δώσατε. Θα ήθελα να πω απλώς ότι έγινε μια σφοδρή συζήτηση στα κοινοτικά θεσμικά όργανα με αντιπαράθεση των διαφόρων απόψεων και ιδεών και διαπιστώνω ότι ο ιδιάζων ρόλος της ανθρωπιστικής βοήθειας έχει γίνει γενικώ αποδεκτός. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι όλοι τελικά καταλαβαίνουν ότι αν εμείς θέλουμε να επιτελέσουμε το έργο μας θα πρέπει να διαχωρίσουμε τη θέση μας από το πολιτικό πρόγραμμα, να είμαστε τελείως αυτόνομοι, γιατί σε πολλές περιοχές του κόσμου επεμβαίνουμε σε ένοπλες συγκρούσεις και αν θέλουμε να σώσουμε ζωές όπως είναι το έργο μας, θα πρέπει να συνεργαζόμαστε με όποια κυβέρνηση μπορούμε, γιατί η πολιτική ή τα διάφορα, οι διάφορες πλευρές ένοπλης σύγκρουσης έχουν διαφορετικές απόψεις και επιθυμίες. Οι, οι φορείς όμως ανθρωπιστικής βοήθειας δεν μπορούν να εμπλακούν στην πολιτική, αλλιώς αλλοιώνουν το έργο τους. Και αυτό το κατάλαβαν και οι υπηρεσίες εξωτερικής δράσης και οι αρμόδιοι για την ανάπτυξη και φυσικά πολύ περισσότερο οι συναδελφοί μου. Τι σημαίνει αυτή η περίφημη περιεκτική προσέγγιση, σφαιρική προσέγγιση. Σημαίνει ότι έχουμε ένα ξεχωριστό ιδιαίτερο καθεστώς όπου αναγνωρίζεται και η ιδιαιτερότητά μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συμμετέχουμε στην ανταλλαγή πληροφοριών ή δεν συμμετέχουμε στη συζήτηση, στην ανάλυση των κινδύνων, στην ανάλυση της τροδότητας της κατάστασης και φυσικά θέλουμε να συμμετέχουμε σε όλα αυτά γιατί είναι προς το συμφέρον μας. Και Ακριβώς επειδή είμαστε πεπισμένοι ότι οι γνώσεις μας για την περίπλοκη εθνοτική κατάσταση στο Νότιο Σουδάν για παράδειγμα μπορεί να χρησιμεύσει και να ενημερώσει καλύτερα τους διαπραγματευτές μας ε, θα καταφέρουμε έτσι να περιορίσουμε τον κίνδυνο μιας ανθρώπινης καταστροφής και χωρί να διακυβεύουμε εδώ την ουδετερότητα και την αμεροληψία μα, θεωρώ ότι έχουμε καθήκον να έχουμε στενή συνεργασία και αγαστή συνεργασία με του συναδέλφου που ασχολούνται με, το πολιτικό σκέλο, με το αναπτυξιακό σκέλο και ούτω καθεξή. Κάτι άλλο που διαπιστώσαμε και χρειάστηκε χρόνο, γιατί χρειάστηκε και εμεί να προσαρμοστούμε, οι εργαζόμενοι στον ανθρωπιστικό κλάδο, το γεγονό ότι είμαστε ανεξάρτητοι και ουδέτεροι αμερόληπτοι δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι δεν θέλουμε καμία επαφή ε, με τις κυβερνήσεις. Σε μερικές περιπτώσεις είναι χρήσιμο να έχουμε διάλογο με τις ε, υγειονομικές αρχές, με τις ε, γεωργικές αρχές, με τις αρχές διαχείρισης του υδατός τους αρμόδιους φορείς ίδρευσης, ώστε να γίνει η καλύτερη πλαισίωση της ανθρωπιστικής βοήθειας με βάση αυτά που γίνονται σε κάθε χώρα. Έχουμε ανοιχτό πνεύμα οι εργαζόμενοι στον ανθρωπιστικό κλάδο. Δεν είμαστε περιχαρακωμένοι στην ανεξαρτησία μας, στην ουδετερότητά μας. Δεν την αναμασούμε ως κανένα θρησκευτικό μάντρα. Γιατί συμμετέχουμε στη δράση επιτόπου και αν έχουμε κυβερνήσεις με σωστή συμπεριφορά, με σωστές ενέργειες, φυσικά και θέλουμε να συνεργαζόμαστε μαζί τους. Κάτι άλλο που θα ήθελα να υπογραμμίσω, το ανέφερα και προηγουμένως στην συζήτηση που είχαμε τον κύριο Γκέρενς για την ε, σύνδεση αναπτυξιακού και ανθρωπιστικού σκέλους. Είναι προφανές ότι οφείλουμε να συνεργαστούμε, να συνεργαζόμαστε με τους συναδέλφους ε, της αναπτυξιακής πολιτικής, ώστε να φροντίσουμε όταν έχουμε μια ανθρωπιστική επιχείρηση σε μια περιοχή ή σε μια χώρα όπου έχουμε ξεπεράσει το πρωταρχικό στάδιο και περνάμε στο δεύτερο στάδιο, όταν ε, αποχωρούμε εμείς να δίνουμε τη σκητάλη στους ε, αρμόδιους για την ανάπτυξη, να υπάρχει κοινό ε, προγραμματισμός, να συνδέσουμε την παροχή βοήθειας, την παροχή ανακούφισης από την έκτακτη ανάγκη με την ε, διευκόλυνση της ανάπτυξης. Έτσι θα ελέγξουμε και καλύτερα τις κρίσεις. Και πιστεύω ότι ως προς το θέμα αυτό, ως προς την ανατροπή αυτή, έχουμε βελτιωθεί και έχει βελτιωθεί και ο διάλογος με τους άλλους φορείς. Πάντως, ε, έχουμε κωδικοποίησει την προσέγγιση μας με πολύ τηλεγραφικό τρόπο έχουμε την περίφημη προσέγγιση ναι μεν μέσα αλλά έξω. In but out. Είμαστε ταυτόχρονα και μέσα και έξω. Δηλαδή συμμετέχουμε στην ανταλλαγή πληροφοριών αλλά δεν δεχόμαστε πολιτικές εντολές και οδηγίες. Παραμένουμε ουδέτεροι σε σχέση με το γενικό πρόγραμμα εργασιών. Ακούμε, δεν είμαστε ανόητοι, ενημερωνόμαστε για τα προγράμματα των ΜΕΝ και των ΔΕ, αλλά οι ανθρωπιστικές δράσεις έχουν στόχο τη διάσωση ζωών και αυτό είναι ο πρωταρχικό στόχο και υπερέχει οποιασδήποτε άλλη προτεραιότητα. Οποιασδήποτε άλλη προτεραιότητα. Φυσικά χρειαζόμαστε καστή συνεργασία, διάλογο και συντονισμό, αλλά θα πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισμός επιτόπου. Και νομίζω ότι είναι πολύ αποτελεσματικός αυτός ο τρόπος εργασίας και έτσι καταφέρουμε να φτάσουμε πραγματικά στις ε, χυμαζόμενες περιοχές από τη συγκρούση, εκεί που υπάρχουν πραγματικά ανάγκες. Ένα άλλο θέμα, μια άλλη πτυχή, όταν μιλούμε για τις επιχειρήσεις επιτόπου, είναι η αγαστή σχέση μεταξύ των αντιπροσωπιών και των γραφείων της ανθρωπιστικής βοήθειας. Θα πρέπει να υπάρχει καλή ανταλλαγή απόψεων επιτόπου. Και υποστηρίζω ένθερμα το ρόλο των επικεφαλής των αντιπροσωπιών, γιατί ήρθατε μια πολιτική ανάλυση πολύ πιο ευρία, έχουν διάλογο με τις κυβερνήσεις, έχουν μια πολύ πιο ευρία προσέγγιση. Από τη στιγμή όμως που μας σέβονται, σέβονται το έργο μας, πιστεύω ότι υπάρχει χώρος για καλή συνεργασία. Και λέω και στους ε, δικούς μου, μην διστάσετε να επισημάνετε τα προβλήματα στους επικεφαλείς των αντιπροσωπιών ή στους συναδέλφους από τον αναπτυξιακό τομέα ώστε να βελτιωθεί η ανάλυση της κατάστασης, ιδιαίτερα στις πιο ευάλωτες χώρες. Κυρία Στρίφλερ, νομίζω ότι σχεδόν εξάντλησα το 7 λεπτό που μου δώσατε και μαζί με τον κύριο Παπόφσκι και τους συναδέλφους ε, ε, που κάθονται δίπλα σα, Έχουμε καταφέρει να βρούμε ένα πεδίο συνεννόηση πολύ επικοδομητικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Ποπόφσκι, θα ήθελα αγαπητοί συνάδελφοι να χαιρετήσω μία αντιπροσωπεία από τους συναδέλφους μας ε, του, της Βουλής της Ιορδανίας. Το πλαίσιο μιας επίσκεψης ε, κοινοβουλίων που οργανώνεται αυτή την εβδομάδα έχουμε πολιτικούς εκπροσώπους αλλά και ε, υψηλά ιστάμενα στελέχη από τη Βουλή της χώρας αυτής. Σας καλωσορίζουμε θερμά στη συνεδρίαση της Επιτροπής μας για την Ανάπτυξη. Και δίνω αμέσως τον λόγο στον κύριο Ποπόφσκι, Γενικό γραμματέα επιτετραμένο σε θέματα ε, ε, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Έχετε 7 λεπτά. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, ένα ερώτημα υπάρχει σε ό,τι αφορά τον τίτλο του πάνελ σε ό,τι αφορά την αρχή της ανθρωπιστικής δράσης και κατά πόσον πρόκειται για κίνδυνο ή για αξία. Κοιτάξτε, αν πιστεύω ότι είναι κίνδυνος δεν θα ήμουν εδώ σήμερα. Θεωρώ λοιπόν ότι πρόκειται σαφέστατα για μια α, προστιθέμενη αξία αυτή η ανθρωπιστική βοήθεια. Φυσικά υπάρχει ένα θέμα όταν ενεργούμε και δρούμε στο εξωτερικό, δρούμε ως πολιτικός φορέας. Δεν είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μια μεγάλη μη κυβερνητική οργάνωση, παρά το γεγονός ότι πολλές φορές έτσι μας αντιλαμβάνονται. Και ξέρουμε ότι η αρχή της ανθρωπιστικής ε, βοήθειας θα πρέπει πάντα να γίνεται σεβαστή ρητά αναφέρεται στην ε, συνθήκη και τα... η συνθήκη λοιπόν θα πρέπει να γίνεται σεβαστή. Αυτή είναι η βάση της συζήτησή μας με τους ομολόγους μας και τους συναδέλφους μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να σας παρουσιάσω λοιπόν ε, ποιο ήταν το ιστορικό της ανακοίνωσης την οποία αναφέρεται και εσείς κυρία Πρόεδρε και ο κύριος Σούτενσεν. Η συζήτηση για την ε, συνεκτική αυτή προσέγγιση δεν είναι ιδιαίτερος καινούρια. Σκοπός μας ήταν να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο πολιτικό που θα αποτυπώνει το πνεύμα και όχι μόνο το γράμμα της συνθήκης της Λισαβόνας και την υποχρέωση για μεγαλύτερη συνεκτικότητα στην εξωτερική μας δράση. Αυτό ακριβώς μας οδήγησε να υποβάλουμε την κοινή αυτή ανακοίνωση, την οποία αναπτύξαμε από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μας πήρε κάποιο χρόνο γιατί είναι περίπλοκη και αγγίζει ευαίσθητα θέματα. Δεν προσπαθώ να το κρύψω αυτό με τα κρατημέλη λοιπόν. Και νιώθουμε ότι η διεθνής κοινότητα ήταν ανυπόμονη όλοι, ήθελαν να δουν επιτέλους την ανακοίνωση αυτή από το Δεκέμβριο. και κατά κάποιο τρόπο πρόκειται για ένα κείμενο κοινή λογική. Ε, να εφαρμοστούν τα μέσα και τα μέτρα που έχουμε στη διάθεσή μας με το βέλτιστο δυνατό τρόπο. Αλλά αυτή η κοινή λογική έχει πλέον ε, μεταφραστεί σε πολιτική, σε μια δήλωση πολιτική που την ε, προσπογράφει και, ο και η Επιτροπή και ο Υπότος Άρμοστης, ο το Εκπρόσωπος Αντί. Η ίδια λοιπόν η ανακοίνωση και η συνεκτική προσέγγιση αναφέρθηκε και από τον Επίτροπο, τον Πρόεδρο Μπαρόζο, στην τελευταίο Συμβούλιο το Δεκέμβριο. Αυτή η έννοια της συνεκτικότητας υπερβαίνει τα θεσμικά όργανα των Βρυξελών. Αν μιλάμε λοιπόν για μια τέτοια προσέγγιση συνεκτική, τι εννοούμε. Να δρούμε από κοινού με συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών. Χρειαζόμαστε λοιπόν και τα κρατημέλη και σε επίπεδο προγραμματισμού της πολιτικής και σε επίπεδο εφαρμογής επιτόπου. Να αναφέρω λοιπόν κάποια, κάποιες κοινέ ε, γραμμές δράσης που αναφέρονται στο κείμενο της ανακοίνωσης. Καταρχάς, μία από κοινού ανάλυση. Εδώ λοιπόν μπορούμε πολύ καλά να συνεργαστούμε με τους ανθρωπιστικούς παράγοντες και το κάνουμε αυτό. Χρειαζόμαστε ένα κοινό όραμα στρατηγικό για κάθε χώρα και κάθε περιφέρεια όπου θέλουμε να δραστηριοποιηθούμε. Πρέπει να τονίσουμε καλύτερα πιο πολύ το θέμα της πρόληψης της συγκρούσεων και να δεσμευόμαστε μακροπρόθεσμα εκ παραλλήλου και μετά να γίνει σύνδεση μεταξύ των διαφόρων πολιτικών σε ό,τι αφορά και τις εσωτερικές πολιτικές αλλά και τις εξωτερικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεταξύ των αντιπροσωπείων με την υπηρεσία εξωτερικής δράσης και λοιπόν πρέπει να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο τους πόρους μας. Το θέμα λοιπόν δεν είναι τόσο πολύ το τι θα πρέπει να κάνουμε, αλλά το πώς θα πρέπει να το πετύχουμε, πώς θα πρέπει να πετύχουμε την καλύτερη στρατηγική συνεκτικότητα σε ό,τι αφορά τα μέσα για την εξωτερική πολιτική. Πολλά από αυτά λοιπόν τα πράγματα, πολλές από αυτές τις ενέργειες τις κάνουμε και τις εφαρμόζουμε εδώ και καιρό. Δεν ε, είναι πραγματικά κάτι καινούριο, αλλά πρόκειται για ένα συνεκτικό πλαίσιο το οποίο θέλουμε πλέον να καθοδηγεί τις δράσεις μας και στην πολιτική ανάπτυξη και στην πολιτική την εξωτερική και την πολιτική άμυνας. Τώρα σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική δράση και το ρόλο της στο πλαίσιο της συνεκτικής προσέγγισης, σύμφωνο απόλυτα με τον κύριο Σούρενσεν. Δεν έχω πολλά να προσθέσω. Μόνο να πω ότι πριν από ένα χρόνο, εγώ και ο Κλάους πήγαμε στο Δουβλίνο, μείναμε μία μέρα για να εξηγήσουμε στην ανθρωπιστική κοινότητα των κριτών μελών ότι δεν υπήρχαν τριβές ή μάλλον υπήρχαν τριβές οι οποίες τελικά οδήγησαν σε ένα αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη του εγγράφου. Και είναι κρίσιμη σημασία να λάβουμε υπόψη την εμπειρία και τη γνώση των ανθρωπιστικών φορέων όταν θέτουμε προτεραιότητες, γιατί πολλά μπορούν να μας διδάξουν. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στο πλαίσιο της πρόληψης συγκρούσεων. Και Πολλοί λοιπόν φορεί μπορούν να διδαχτούν και πολλά από τους ανθρωπιστικούς φορεί σε ό,τι αφορά την ε, ευελιξία και την ταχύτητα. Εδώ θα πρέπει να κάνουμε μεγάλη προσπάθεια και προσπαθούμε λοιπόν να, λοιπόν, να εμπνευστούμε από τον τρόπο που δράτε. Παρά το γεγονό που έχουμε, ότι έχουμε περιορισμούς. Κατά δεύτερον, το πώ ε, είναι η επικοινωνία με τα κράτη-μέλη. Και τέλο, αλλά εξίσου σημαντικό, η παράδοση της ανθρωπιστικής κοινότητας να δραστηριοποιείται επί τόπου με τους τοπικούς φορείς και να χρησιμοποιεί τη γνώση των τοπικών φορέων, των μη κυβερνητικών οργανώσεων για παράδειγμα. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό το μάθημα λοιπόν και θα πρέπει να αποτελεί τη βάση μιας πραγματικά συνεκτικής προσέγγισης. Φυσικά, έπειτα και συνέχεια θα πρέπει να γνωρίσουμε τις διάφορες ε, περιοχές να ξεπεράσουμε κάποιες ευαισθησίες, το φόβο ίσως ο ένας του άλλου. Θα πρέπει να εξηγούμε, ιδιαίτερα σε άτομα που έχουν ε, θέμα με την ασφάλεια, ότι έχουμε ειρηνικούς σκοπούς και ότι δεν σκοπεύουμε να αναμειχθούμε σε συγκρούσεις. Και να παραθέσω και ένα παράδειγμα κλείνοντας, γιατί πριν από κάποιες ώρες ε, οι Υπουργοί Εξωτερικών έλαβαν μία απόφαση να ξεκινήσουν λοιπόν μία αποστολή ε, ΚΕΠΑ στην Κεντρική Αφρική. Ξεκινάει λοιπόν ο προγραμματισμός, ο λειτουργικός, ε, επιχειρησιακός ε, προγραμματισμός. Ήταν λοιπόν η ανθρωπιστική κοινότητα που κρύβεται πίσω από αυτή την απόφαση, γιατί λάβαμε μεγάλη ενθάρρυνση και από τους συναδέλφους και η Επίτροπος και ο κύριος Μπαρόσο, αλλά και από την ΟΗΕ. Όλοι λοιπόν από εμά περίμεναν να λάβουμε την απόφαση να δραστηριοποιηθούμε. Αυτό λοιπόν και συνέβη. Αυτή είναι λοιπόν η προστιθέμενη αξία και ειλικρινά ακτιμώ ότι το θέμα της ανθρωπιστικής, ε, των ανθρωπιστικών ε, φορέων ίσως να έχει υπερεκτιμηθεί. Δεν νομίζω ότι έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα. Καταλαβαίνουμε ένα τον άλλον και άλλωστε έχουμε και τους ίδιους στόχους Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στην κυρία Κατρίν Σίκε για 7 λεπτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία αυτή να σας παρουσιάσουμε και την ε, πλευρά των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Νομίζω ότι παρακολουθήσαμε την εξέλιξη της ανακοίνωση από κοντά, εκτός του και χαιρόμαστε που επιτέλους την βλέπουμε Χαιρόμαστε που βασίζεται σε συνένεση καταρχάς. Νομίζω ότι αυτό αποτελεί μια πολύ θετική ένδειξη. Επικεντρώνεται στον κοινό προγραμματισμό και καταρχάς στην πρόληψη των συγκρούσεων. Αυτό είναι λοιπόν πολύ θετικό. Το ότι πλέον το έχουμε σε χαρτί, ότι αυτή θα πρέπει να είναι η κινητήριος δύναμη πίσω από την συνεκτική προσέγγιση. Αναφέρεται η κοινωνία των πολιτών πλέον και ότι κάθε κρίση είναι διαφορετική. Άρα η αντιμετώπιση θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στην κρίση σε ό,τι αφορά τη συνεκτική προσέγγιση. Κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ο πλήρης σεβασμός και η εντολή να γίνεται σεβαστή η εντολή του κάθε φορέα. Το ανέφερε και ο προλαλή σα. Αυτό αναφέρεται και στη συνθήκη. Όλα αυτά λοιπόν είναι τα θετικά στοιχεία. Το θέμα λοιπόν είναι, όπως πάντα, πώς εφαρμόζονται όλα αυτά τα θετικά στοιχεία. Εδώ λοιπόν είναι η πρόκληση. Αυτό άλλωστε το είδαμε Νομίζω ότι αυτές οι αρχές ε, μας βρίσκουν σύμφωνους όλους τα τελευταία δύο-τρία χρόνια. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε και πιο πολύ επ' αυτών. Το θέμα είναι πώς εφαρμόζονται όλα αυτά στην πράξη. Από την ανακοίνωση μέχρι τις επιχειρήσεις επιτόπου. Να αναφέρω λοιπόν κάποια σημεία όπου θεωρώ ότι υπάρχουν και ελοχεύουν προκλήσεις και κίνδυνοι για όλους τους φορείς σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της ε, ανακοίνωσης. Καταρχάς υπάρχει έντονη σύνδεση μεταξύ της ανάπτυξης και της ασφάλειας. Όταν συνδέει κανείς ε, τι τις ανθρωπιστικές δράσεις και την ασφάλεια, το αποτέλεσμα είναι διαφορετικό, ξέρετε. Για μας η ασφάλεια είναι βάση προκειμένου να υπάρχει πρόσβαση στον κόσμο και να μπορούμε να δρούμε επί Και νομίζω ότι το παράδειγμα το οποίο μόλις αναφέρετε ήταν σαφέστατο. Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Η ανάπτυξη είναι πιο πολιτική φύσεω. Κάτι άλλο, όταν αναλύουμε τις ε, ανάγκες που υπάρχουν, όταν αναλύουμε από κοινού μια κρίση και τα κράτη τα οποία θέλουμε να υποστηρίξουμε, υπάρχει το ερώτημα το κατά πόσον ε, είναι οι ίδιες οι ανθρωπιστικές ανάγκες και οι ανάγκες σε ό,τι αφορά την ε, ασφάλεια. Ενδεχομένως ναι, ενδεχομένως και όχι, θεωρώ. Ένα άλλο ζήτημα. Αν θέλουμε να ενισχύσουμε πιο πολύ την ε, επιχειρησιακή συνεργασία, υπάρχουν πάρα πολλοί θετικέ συνεργασίες και η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστική Βοήθειας έχει ε, συμμετάσχει σε πολλές δράσεις και ο Ερυθρό Σταυρό. Αλλά η επιχειρησιακή συνεργασία θα πρέπει επίσης να έχει πολύ σαφή ορισμό. Γιατί αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε με το βέλτιστο τρόπο τα εργαλεία και τα μέσα που έχουμε, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τότε η καλύτερη και η βελτιστή χρήση της ανθρωπιστικής βοήθειας είναι να σέβεται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων όπως διαμορφώνονται τα τελευταία 20 χρόνια. Ένα ακόμα ζήτημα το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι σημαντικό να υπάρχει μια γεφύρωση με την ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να υπάρχει βιώσιμη λύση. Και εμείς ε, με το θέμα της ε, ανοχής, όχι μόνο της πολιτικής, αλλά και της κοινωνικής. Η πολιτική λοιπόν αυτή ανοχή έχει να κάνει με την ε, ε, τρομοκρατία, την στρατιωτική παρέμβαση και με την εσωτερική ασφάλεια ασφαλώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν νομίζω ότι μια συνεκτική προσέγγιση καταρχάς μπορεί να δημιουργηθεί για να είναι αλτρουιστική στη φύση της και τη λειτουργία της σε όλο τον κόσμο. Όχι, έχουμε ένα σαφή στόχο τον οποίο και εξυπηρετούμε. Τώρα, να αναφέρω κάποιες συστάσεις. Πολύ σημαντικές θεωρώ για να παρακολουθούμε το πόσο αυτά εφαρμόζονται, γιατί μου έκανε εντύπωση που αναφέρεται ρητά στην ε, ανακοίνωση ότι όλοι οι φορείς της Βρυξέλλες, όχι μόνο στα θεσμικά όργανα πρέπει να βρουν. Θεωρώ λοιπόν ότι χρειάζεται μια καλή πολιτική ε, ενημέρωσης. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ενημέρωση και η επικοινωνία σε ό,τι αφορά ε, τη δημιουργία κάποιων κοινών αρχών και μια κοινή νοτροπίας και είναι πολύ εύκολο να θολώσουν τα νερά. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα τα τελευταία χρόνια όπου δεν ήταν σαφές κατά πόσο η ανθρωπιστική βοήθεια ήταν τμήμα της συνεκτική προσέγγιση ή όχι. Αυτό λοιπόν θα είναι ενδιαφέρον να το δούμε για το μέλλον. Κάτι άλλο σε ό,τι αφορά τον συντονισμό και τον προγραμματισμό. Η πλατφόρμα για, την κρίση, για τις κρίσεις λειτουργεί όλο και καλύτερα. Αποτελεί μια πολύ καλή πλατφόρμα και θα λειτουργεί όλο και καλύτερα στο μέλλον. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις επαφές με την κοινωνία των πολιτών, νομίζω ότι, ότι και αυτό έχει να κάνει ιδιαίτερως με την πρόληψη των συγκρούσεων. Θα ήταν λοιπόν ενδιαφέρον να δούμε ποιοι μηχανισμοί θα χρησιμοποιηθούν και θα υπάρξουν και στις Βρυξέλλες αλλά και επιτόπου Και χάρηκα με αυτά που αναφέρατε σε ό,τι αφορά την κοινωνία των πολιτών επίτόπου τόπου στο Νότο. Δυστυχώς όμως αυτό δεν αναφέρεται ρητά στην ανακοίνωση. Ένα επιπρόσθετο στοιχείο, το θέμα του μνημονίου κατανόησης Ω εργαλεία μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμα, αλλά ενδεχομένως και κενά νοήματος τέτοια μνημόνια. Σε κάποιες περιπτώσεις ε, αρμόζει μία λύση και σε κάποιες άλλες όχι. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα μνημόνια αυτά κατανόησης, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να κατανοήσουμε ότι εκεί αναφέρονται οι σαφείς ρόλοι και οι σαφείς εντολές και η συμπληρωματικότητα των διαφόρων φορέων στους ε, διάφορους ε, μηχανισμούς. Έχουμε ανθρωπιστική βοήθεια, έχουμε την προστασία των πολιτών, έχουμε το στρατό, όλα πολύ ε, ισχυρά εργαλεία και θα πρέπει να υπάρχει συμπληρωματικότητα. Αυτή η συμπληρωματικότητα λοιπόν σε διεθνέ επίπεδο είναι μια πρόκληση και τα αρχικά μνημόνια κατανόηση. Θυμάμαι ότι υπάρχει μια μεταξύ τη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη Εξωτερική ε, Υπηρεσία Εξωτερική Δράση σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική δράση. Θα είναι λοιπόν πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί μας πήρε πάρα πολύ χρόνο να την αναπτύξουμε. Έχουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε και κάποιες προκλήσεις στο μέλλον. Και το ερώτημα λοιπόν είναι πότε μπορεί κανείς να ανακηρύξει μια χώρα για το ότι χρήζει ε, κοινή ανάλυση, τέτοια συνεκτική ανάλυση. Είδα ότι υπάρχουν κάποια συστήματα έγκυρη προειδοποίηση. Κοιτάξτε, εγώ μόλις 50 είμαι, αλλά έχω την ε, ελαφρά εντύπωση ότι μας δίδονται επαρκείς ενδείξεις και ε, επαρκείς ε, προειδοποιήσεις για κρίσεις Επί μακρόν, Το θέμα είναι η πολιτική βούληση να αναπτυχθεί κάτι. Και αυτό που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια είναι το εξή. Ότι αυτό πάντα καθυστερεί. Και τότε όλοι αναγκαζόμαστε να καταβάλουμε μεγαλύτερε προσπάθειε. Εδώ θα ήθελα να κλείσω και να σα δώσω το χρόνο να μου πείτε και τις δικές, να μα αναφέρετε και τι δικέ σα σκέψει. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ. Κατρίνα, δώσω τώρα το λόγο στον Αντών Ζεράρ, που είναι υποδιευθυντή του Τμήματο Συντονισμού και Απόκριση τη ΟΝΟΤΣΑ για 7 λεπτά. Κύριε Ζεράρ. Ευχαριστώ, κύριε Στίφλερ. Και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση του γραφείου, ιδιαίτερα για, την, για το συντονισμό και την απόκριση. Ε, είμαστε κάπως outsiders σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θα ήθελα να σας ε, δώσω και το πρίσμα των συνομιλιών όχι μόνο με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και με το ΝΑΤΟ που είχε πριν από λίγο καιρό μία διάσκεψη για το θέμα αυτό. Και στο ΝΑΤΟ λοιπόν γίνονται τέτοιες συζητήσεις για το κατά πόσο στην προσέγγιση θα πρέπει να λαμβάνεται και η ανθρωπιστική διάσταση. Αυτή η περιεκτική προσέγγιση, η σφαιρική προσέγγιση έχει γίνει η πολύ συνηθισμένη έκφραση σε πολλά κοινωτικά και άλλα θεσμικά όργανα και περιγράφεται μια νέα διοργανική προσέγγιση που πρέπει να περιλαμβάνει περισσότερους, όπως είπε ο κ. Ποπόφσκι, πρέπει να είναι πιο συνεκτική, πιο συντονισμένη. Ταυτόχρονα είδα εκατοντάδες διαφορετικούς ορισμούς αυτής της σφαιρικής προσέγγισης. Απρός global, το λέμε στα γαλλικά, εφαρμόζουμε διαφορετικό τρόπο. Ε, και το ίδιο πολύ διαφορετικά θα ε, το ερμηνεύσει η Βρετανική κυβέρνηση, η Καναδέζικη και ούτω καθεξής. Οπότε θα πρέπει να είμαστε κάπως πιο σαφείς για το τι εννοούμε όταν λέμε περιεκτική προσέγγιση ή σφαιρική προσέγγιση. Να κάνουμε και κάποια σχόλια για αυτή τη νέα ανακοίνωση και χαίρομαι για την κοινή ανακοίνωση περί περιεκτικής προσέγγισης ε, και την επιθυμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για καλύτερα συντονισμένη στρατηγική αποτελεσματική εξωτερική δράση. Πάνω απ' όλα όμως στο γραφείο μας ε, στα Ηνωμένα Έθνη για το συντονισμό και την απόκριση μας ενδιαφέρει ε, η ιδιαίτερη αναγνώριση της ανθρωπιστικής βοήθειας στην κοινή ανακοίνωση και χαίρομαι που αναφέρονται οι ανθρωπιστικές αρχές και η, η Ευρωπαϊκή Συνένεση για τα ανθρωπιστικά θέματα, όπω είπαν οι συνάδελφοι. Γιατί όμω είναι τόσο σημαντικό να γίνονται αυτέ οι μνήε επισήμω στι ε, ανακοινώσει. Εξορισμού, η περιεκτική προσέγγιση είναι εξορισμού ε, πολιτική. Εδράζεται στο πολιτικό θεματολόγιο και στο πολιτικό όραμα είτε χωρών είτε οργανώσεων. Σήμερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από δύο χρόνια του ΝΑΤΟ. Μια και το γραφείο μας ε, είναι επιφορτισμένο με το συντονισμό της ανθρωπιστικής δράσης, μας απασχολεί κάπως ότι οι ανθρωπιστικοί φορείς θα ενταχθούν στο τμήμα μιας πολιτικής περιεκτικής ή προσέγγιση. προσέγγισης. Είτε στα πλαίσια μιας λειτουργίας, είτε στα πλαίσια μιας ανακοίνωσης. Εμείς προωθούμε τις ανθρωπιστικές δράσεις και όταν δεν θέλει κανείς να, συλλάβει, να συμβάλλει σε πολιτική προσέγγιση, ίσως δημιουργηθεί μια ασφαλμένη ε, εντύπωση. Και η πλήρης ένταξη της ανθρωπιστικών φορέων ε, σε, στη διαχείριση κρίσεων ίσως τους οδηγήσει σε μια αναποτελεσματική δράση, κάτι που θα ε, προκαλέσει αρνητικέ συνέπειες. Γιατί αν συμπεριληφθούν στην περιεκτική προσέγγιση τα ανθρωπιστικά επιτεύγματα και ανθρωπιστικές ε, διαπραγματεύσεις, θα παρεμποδιστεί η δράση τη αμερόληπτη και ανεξάρτητης δράση τη ανθρωπιστική ενέργεια. Γιατί για την ανθρωπιστική ενέργεια θα πρέπει να γίνεται αναγνώριση τη από του πάντε και να μην θεωρηθεί η, αναγνωριστική, η ανθρωπιστική βοήθεια ω τμήμα τη πολιτική δράση. Και αν θέλουμε να φτάσουμε αποτελεσματικά στους πληθυσμούς ε, σε ένοπλε συγκρούσει και στι τοπικέ κοινότητε ή άλλου φορεί, θα πρέπει να αποδεχθούμε και εμεί και αυτοί το ρόλο των ανθρωπιστικών φορέων ως ουδέτερων, αμερόληπτων φορέων ανθρωπιστικής βοήθειας. Γι' αυτό και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ε, την ε, σταθερή ε, προσήλωση στις βασικές αρχές. Και η έννοια αυτή της αντίληψης είναι δυσνόητη, γιατί αν μία πλευρά σωστά ή λάθος θεωρεί ότι οι ανθρωπιστικοί φορείς εξυπηρετούν μία συγκεκριμένη πολιτική έκβαση και ότι δεν εφαρμόζεται η ανθρωπιστική δράση μόνο για ανθρωπιστικές ανάγκες, τότε κατά πάσα πιθανότητα η πλευρά αυτή δεν θα επιτρέψει την ανάπτυξη των ανθρωπιστικών δραστηριοτήτων. Η UNOCHA με βάση τη λειτουργία της έχει ιδιαίτερο καθήκον όχι μόνο να προωθεί την, το συντονισμό σε ανθρωπιστικά θέματα αλλά να έχει πολύ προσεκτική επαφή με άλλα τμήματα του, της Γενικής Γραμματείας και κυρίως με πολιτικούς φορείς ή άλλους γιατί τα Ηνωμένα Έθνη ως, πολιτικό, ως πολιτική οργάνωση θα πρέπει να εξασφαλίσει την εφαρμογή ε, ολοκληρωμένων ε, αποστολών και να παρόλα αυτά να σεβαστεί την ανεξαρτησία των ανθρωπιστικών φορέων και οργανώσεων. Γιατί εμείς ε, θεωρούμε ότι η προσέγγιση μας είναι περισσότερο συμβουλευτική σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκέλος, το σκέλος εδραίωσης της ειρήνης και όχι ως περιεκτική. Και οι, οι συνδυασμένες αποστολές στηρίζονται στην εντολή του ΟΗΕ που καθορίζει σαφώς το ρόλο των διαφόρων φορέων μετά από εξονυχιστική ανάλυση. Δεν είναι ένα θεσμικό θεματολόγιο, αλλά κάνει σαφή διαχωρισμό. Επίση, οι ολοκληρωμένε αποστολέ επιτρέπει στους ανθρωπιστικού ε, παράγοντε να μένουν εκτό τη ε, ολοκληρωμένη αποστολή. Όταν μια πολιτική αποστολή ή εδραίωση ειρήνης ε, αναπτύσσεται σε περιοχές μεγάλης αστάθειας όπως τον Ταρφούρη, η εδραιωση ειρηνης αναπτυσσεται σε περιοχες μεγάλη ασταθειας όπω τον Νταρφούρι, η σομαλια το Γραφείο για το Συντονισμό Ανθρωπιστικών Θεμάτων και άλλοι ανθρωπιστικοί φορεί θα μείνουν σαφώς διαχωρισμένοι από την δομή της αποστολής για να εξασφαλιστεί η ιδιωτερότητά τους και να μπορούν να παρέχουν τις ανθρωπιστικές δραστηριότητες και να σώζουν ζωές. Σε ό,τι αφορά το τμήμα του ΟΗΕ για την εδραίωση της ειρήνης, γνωρίζουμε ότι η υποχρεωτική ολοκλήρωση εκεί που δεν είναι απαραίτητη, ίσως είναι αναποτελεσματική και αντιπαραγωγική. Οπότε μας ενδιαφέρει το συνολικό υπόβαθρο μας ενδιαφέρει η διαφάνεια του πολιτικού και στρατικού θεμελιωγίου, ο σεβασμός των ε, εντολών και επίσης αφής επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Όλα αυτά έχουν σημασία. Οπότε μια οργάνωση όπως τα Ηνωμένα Έθνη και με την υποστήριξη Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την ε, ε, διεκπαιρέωση των εντολών μας. Έχουμε ταυτόχρονα εντολή ως φορείς ανθρωπιστικής ενέργειας να ανακουφίσουμε τον ανθρώπινο πόνο και τις οδύνες και την οδύνη στον Παγκουή, στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, στον Νότιο Σουδάν ή αλλού. Και γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε υγιείς και απόμακρες σχέσεις από τους πολιτικούς φορείς και να τηρήσουμε τους στόχους της δικής μας οργάνωσης. Οπότε κοινή ανακοίνωση που αναγνωρίζει αυτή την ιδιαιτερότητα της ανθρωπιστικής αποστολής ε, είναι πολύ σημαντική. Βέβαια η ανακοίνωση αυτή, όπως είπε και η συνάδελφη αυτή τη Voice, αφήνει μεγάλο περιθώριο ε, για την ε, διακριτική ευχαίρεια της εφαρμογής και του ορισμού της περιεκτικής προσέγγισης. Θα πρέπει η ενισχυμένη συνεργασία να μην αποβεί βάρος του ανθρωπιστικού προγράμματος, ιδιαίτερα στα πλαίσια των δράσεων εκτάκτου ανάγκης. Γι' αυτό και θα έλεγα να ε, προσέξουμε ιδιαίτερα στο θέμα της εφαρμογής αυτής της ε, ε, περιεκτικής προσέγγισης, σφαιρικής προσέγγισης. Σας ευχαριστώ. Ήταν εκπληκτικές και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες οι ομιλίες σας. Θα έχουμε τώρα ένα χρόνο, λίγο χρόνο για τις ερωτήσεις και τη συζήτηση. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Γκέρενς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους ε, ομιλητές διότι μας ε, διαφώτισαν. Καταλάβαμε καλύτερα τις διάφορες αποχρώσεις έννοιες του όλου θέματος που μας απασχολεί. Ήμουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 1995 όταν γινόταν λόγος για την πρόληψη της γενοκτονίας στην Ρουάντα και συνεχώς λέγαμε ότι ε, πρέπει να δοθούν προειδοποιήσεις και τα λοιπά, ε, ότι θα είχαμε προειδοποιητικές ενδείξεις, ενώ όλοι το ήξεραν τελικά. Ερωτώ λοιπόν σήμερα με τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα μαθήματα που ελπίζω ότι πράγματι έχουν μάθει ε, τα Ηνωμένα Έθνη και οι λοιποί θεσμοί ε, μετά την αποτυχία της δεκαετίας του 90 στην Ρουάντα. Μετά από όλα αυτά λοιπόν ε, έχει πραγματικά εξαλειφθεί αυτό το ενδεχόμενο πλήρους αποτυχίας. Ε, μπορεί να ξαναυπάρξει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Τι μπορούμε να ελπίζουμε. Αυτό είναι το ερώτημά Εξαιρετικό το ερώτημα. Δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Έτσι δεν είναι. Α, ο κύριος Κορτές Λάστρα, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές για τις πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες τους. Μάθαμε πολλά. Ακολουθώ λοιπόν τη γραμμή που παρουσίασε ο κύριος Γκέρετς, γιατί θέλω να σχολιάσω και να πω το εξής. Μιλούμε για την ανθρωπιστική βοήθεια. Καλώς. Ενίοτε όμως το συνδέουμε και μιλούμε για ανθρωπιστική παρέμβαση. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, όταν κάνουμε αυτή την ανθρωπιστική παρέμβαση, τελικά ε, δυσκολευόμαστε στη συνέχεια να το αποσυνδέσουμε από την πολιτική μας δράση, γιατί ανθρωπιστική δράση είναι αυτή η, την οποία θέλουμε να κάνουμε, έτσι δεν είναι, και έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το οποίο είπε ο κ. Ζεγάχ, δηλαδή πρέπει να διανύσουμε μεγάλη απόσταση, να μιλήσουμε με όλους τους συνομιλητές μας επιτόπου, έτσι ώστε να καταστήσουμε σαφές ότι άλλο πράγμα είναι η δική μας ανθρωπιστική βοήθεια και άλλες είναι οι ανθρωπιστικές παρεμβάσεις, το δικαίωμα παρέμβασης, η ευθύνη προστασίας την οποία υπομιζόμαστε και η ευθύνη ε, παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας σε εκατομμύρια ή σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Ήθελα λοιπόν να μοιραστώ μαζί σας αυτό τον προβληματισμό, διότι τον θεωρώ σημαντικό και σύν της άλλη συμφωνώ με τον κύριο Ζεράρ ε, σε σχέση με τη συνολική προσέγγιση, το συνολικό σημείο εστίασης το οποίο ε, τόνισε στο μέλλον δεν θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε για θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας χωρίς την ύπαρξη ασφάλειας. Αυτό πάει χέρι με χέρι από τη μία, από την άλλη είναι πολύ δύσκολο να δούμε ξεκάθαρα τις διαφορές μεταξύ των δύο. Πώς μπορούμε να τα βελτιώσουμε λοιπόν αυτά για να έχουμε πιο ξεκάθαρο πεδίο δράσης στο περιθώριο των ανθρωπιστικών μας παρεμβάσεων. Ευχαριστώ πολύ. Η Πρόεδρος. Και εγώ σας ευχαριστώ. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να δώσω το λόγο στους ομιλητές του πάνελ. Ποιος θέλει να απαντήσει, ε, υπάρχει κάποιος που να θέλει να απαντήσει, όπως νομίζετε, με τη σειρά που επιθυμείτε εσείς. Ποιος ξεκινάει. Ή να αποφασίσω εγώ. Καλώς, ο κύριος Σόρενσεν. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Σόρενσεν. Θα ακολουθήσω το κατάλογο που έχω μπροστά μου. Ναι, λέει ο κύριος Σόρενσεν, αλλά κοιτάξατε από την άλλη πλευρά. Ήσασταν από αυτή την πλευρά προηγουμένως, κύριε Σόνεσε, γι' αυτό. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερος διότι βλέπω ότι έχουμε εκπροσώπους από το Κοινοβούλιο της Ιορδανίας. Διανύεται πολύ δύσκολες στιγμές. Σας έχουμε στο μυαλό μας, σας σκεφτόμαστε. Είμαστε δίπλα σας, χαιρόμαστε που είστε εδώ και ελπίζουμε ότι θα είναι καλά τα νέα τις επόμενες ημέρες και μήνες. Αυτό καταρχάς. Κατά δεύτερο λόγο, για όλα αυτά τα θέματα, ξέρετε, έχουμε την εξή έκφραση στα αγγλικά που λέει ότι κανείς δεν μπορεί να ξέρει μια πουτίνγκα αν είναι γευστική εκτός και αν τη δοκιμάσει. Εννοώ δηλαδή με αυτό ότι στην καθημερινή πρακτική θα δούμε εάν τα πράγματα λειτουργούν ή όχι. Εγώ δεν ανήκω σε αυτούς που ε, συνεχώς συγγράφουν κείμενα για ενδυνάμιση κρούσης και ούτω καθεξής. Βεβαίως όλα αυτά είναι υποσυζήτηση. Εάν η διαφωνία είναι για το ποια θα αεροσκάφη θα χρησιμοποιηθούν για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας, βεβαίως αυτό συζητείται για το ποιο θα μπει σε αυτέ τι πτήσει τη ΕΚΟ, τη ανθρωπιστική βοήθεια, τότε εγώ βεβαίω συμφωνώ ότι δεν θέλω κανεί πολιτικό ή στρατιωτικό να μπει σε μια τέτοια πτήση για οποιοδήποτε λόγο. Είναι πολλά ζητήματα δηλαδή που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα. Βεβαίω συμφωνούμε όλοι για τη συνολική προσέγγιση, για το να περπατούμε χέρι με χέρι, αλλά η κάθε κατάσταση είναι διαφορετική και θα πρέπει να αναλυθεί το θέμα αναπερίπτωση. Ο Αντουάν Ζεγάχ μίλησε για τι ε, ενοποιημένε αποστολέ στο σύστημα σύστημα των Ηνωμένων Εθνών. Σίγουρα, Αντουάν, συμφωνείτε μαζί μου, η συζήτηση είναι αρκετή αρκετά έντονη μεταξύ του Γραφείου Ανθρωπιστικής Βοήθειας των ΗΠΑ Εθνών, του DPKO και διαφόρων άλλων φορέων. Ε, δίνουμε μάχη για να διατηρήσουμε την ανεξαρτησία μας, ενώ συνάμα θα ε, εγγυόμαστε την ασφάλεια του προσωπικού. Βεβαίως και τη χρειαζόμαστε και δεν χαίρομαι ιδιαίτερως με την ενοποιημένη αποστολή στη Σομαλία. Νομίζω ότι η γλώσσα που υιοθετήθηκε ήταν κάπως υπερβολική ε, στο θέμα της Σομαλίας. Προσπάθησε να το προλάβω, δεν τα κατάφερα, ούτε ο Αντουάν θα μπορούσε να το είχε προλάβει. Να είμαστε ειλικρινείς, δηλαδή είναι μια μάχη που δίνουμε καθημερινά με πολλές μικρές νίκες καθημερινά ή όχι. Από εκεί και πέρα, ναι, ε, Κάθριν, πιστεύω ότι πρέπει να βελτιώσουμε το ραντάρ μας εντός εισαγωγικών που θα προβλέπει και θα προλαμβάνει τις καταστροφές. Καλό είναι το ερώτημα. Είμαστε σήμερα καλύτεροι από ό,τι ήμασταν στην εποχή της Ρουάντα. Ναι, αλλά δεν μπορώ να εγγυηθώ βεβαίως ότι αυτό δεν θα ξανασυμβεί ποτέ. Με την πάροδο των ετών, με την αυξημένη από κοινού χρησιμοποίηση ε, πληροφοριών και στοιχείων σίγουρα θα βελτιωθούμε. Δεν ήμασταν εξαιρετικά καλοί ούτε στο Μαλί, ούτε στο Νότιο Σουδάν, ούτε στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, αλλά γενικότερη βούληση είναι να προχωρήσουμε προ τα εμπρό Η επίτροπο Κρυσταλίνα Γεωργίευα πήγε στην Κεντροαφρικανική ε, Δημοκρατία από πολύ νωρί και προσπάθησε να ασκήσει ε, προληπτική διπλωματία. Έχουμε και το θέμα της Νιγηρίας. Ε, πού θα προκύψει το επόμενο ατύχημα δεν το γνωρίζω. Ωστόσο έχουμε περισσότερα και καλύτερα εργαλεία από ό,τι είχαμε πριν από πέντε χρόνια. Ελπίζω λοιπόν ότι με αυτά τα ψήγματα απάντησης κατάφερα κύριε Γκέρενς να σας δώσω κάποια ελπίδα. Τέλος, ένα θέλω να πω, το εξής. Αυτό που βοηθά ιδιαιτέρως σε αυτή την τόσο περίπλοκη συζήτηση είναι το εξής θα πρέπει ο κάθε λειτουργός, ο κάθε φορέας να ε, τηρήσει ε, την εντολή που του έχει δοθεί. Το πρόβλημα δημιουργείται και περιπλέκεται όταν εγώ, για παράδειγμα, προσπαθήσω να κάνω διπλωματική δουλειά και οι διπλωμάτες προσπαθήσουν να κάνουν ανθρωπιστική δουλειά. Να κάνω εγώ διπλωματική δουλειά μόνο σε αγαστή συνεργασία με τους διπλωμάτες και αντιστρόφως. Το ίδιο και με τους στρατιωτικούς. Εμείνατε στην εντολή σας. Αν χειρίζεστε εσείς καλύτερα τα όπλα και τις επιχειρήσεις ασφαλείας, αυτό να κάνετε και αφήστε μας ήσυχους. Και βεβαίως μπορούμε να συνεργαστούμε και να ανταλλάξουμε πληροφορίες. Αυτό είναι εφικτό. Η Πρόεδρος. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Ποπόφσκι τώρα. Σας ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω με την εφαρμογή του follow-up. Φυσικά θα πρέπει να λειτουργήσει, αλλά αυτό δεν πρόκειται να συμβεί σε μία νύχτα και όπω αναφέρθηκε, υπάρχουν κάποιες τριβέ, κάποιες εντάσει που θα πρέπει να ξεπεράσουμε το βλέπω και εγώ όταν ε, προγραμμάτιζα να πάω στην, ε, στο Κονγκό και μου είπαν ότι ε, με περιορίσαν σε ό,τι αφορά τις πτήσεις μου. Αυτό, εντάξει, δεν θα πρέπει να υπερβάλλουμε και με τα θέματα αυτά. Εδώ είμαστε για να τα επιλύσουμε. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σαφής ο ρόλος της ανθρωπιστικής κοινωνίας. Η συμμετοχή σε κάτι δεν σημαίνει ότι θα τα παίρνουμε όλα αυτά από έναν. Συμμετέχουμε λοιπόν σε μια επιχείρηση. Δεν συμμετέχουμε στην πολιτική, στη στρατιωτική αποστολή. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι κεκτημένο, πώς να σας πω. Αλλά οι ανθρωπιστικοί φορείς μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Ε, για παράδειγμα, αναφέρθηκε αυτή η ανθρωπιστική όθηση για να δραστηριοποιηθούμε στην κεντροαφρενικανική δημοκρατία. Αλλά αυτό δεν έγινε στην Λιβύη, για παράδειγμα η ανθρωπιστική κοινότητα μας προειδοποίησε εκεί να περιμένουμε και να μην αναμειχθούμε. Αυτό και πράξαμε. Νομίζω λοιπόν ότι επί αυτής της βάσης μπορούμε να συνεχίσουμε. Η εμπειρία του ΟΙΕ. Εγώ βλέπω από αυτά που κάνω με τον ΟΙΕ ότι υπάρχει σαφές ενδιαφέρον να δραστηριοποιηθούν πολλά, πολλές υπηρεσίες του ΟΙΕ Είμαι μέλο τη επιτροπή τη Κοινής Επιτροπής ΟΗΕ και Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση κρίσεων. Ξεκίνησε ε, ως ε, ε συμφωνία μεταξύ Υπηρεσία εξωτερική δράση και σώματο του ΟΗΕ. Τώρα πλέον όμως συμμετέχουν πολλοί φορείς του ΟΗΕ και αυτό είναι πολύ σωστό. Όλοι θέλουν να συνεισφέρουν στην πλατφόρμα αυτή για την αντιμετώπιση των κρίσεων που αναφέρθηκε. Σε ό,τι αφορά το σκέλος της πρόληψης, φυσικά θέλουμε να είμαστε καλύτερα εξοπλισμένοι. Θέλουμε να είμαστε σε καλύτερη θέση να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση επιτόπου. Έχουμε ξεκινήσει ένα πιλωτικό πρόγραμμα στο Σαχέλ και θα το επεκτείνουμε. Αλλά Νομίζω ότι όλοι έχουμε διδαχθεί από την περίπτωση της Ρουάντα. Νομίζω ότι η εμπειρία της Ρουάντα έχει ε, καθορίσει και την αρχή της ε, ευθύνης για προστασία, κάτι στο οποίο προσυπογράφουμε. Αλλά συγκεκριμένα για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Χρησιμοποιήθηκε ο όρος γενοκτονία από τον ΟΗΕ όταν συζητήσαμε πρώτο το θέμα αυτό της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας κάποια στιγμή πέρσι τον Οκτώβριο-Νοέμβριο. Ε, επιβεβαιώθηκε και καταφέραμε να επιταχύνουμε την όλη διαδικασία για να φτάσουμε στην σημερινή απόφαση που είναι πολύ σημαντική και ευπρόσδεκτη από τους ανθρωπιστικούς φορείς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ΟΗΕ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο κυρία Σίκ. Λίγα σύντομα σχόλια. Χαίρομαι που ανακύπτει και πάλι το θέμα της ανάγκης ο κάθε φορέας να εμένει στην αντολή του και να περιορίζεται από αυτήν γιατί το θέμα αυτό είναι στην επικαιρότητα εδώ και 4-5 χρόνια και εξακολουθεί να έχει σημασία. Κύριε Κόρτες, δώσατε το χαρακτηριστικό παράδειγμα της σύγχυσης στην επικοινωνία. Γιατί όταν μιλούμε για ανθρωπιστικές δράσεις και για ανθρωπιστική παρέμβαση, θα πρέπει να κάνουμε διαχωρισμό γιατί μπορεί την ορολογία να την ξέρουμε οι ειδικοί, αλλά ο απλός άνθρωπος δεν καταλαβαίνει. Μερικές φορές έχουμε ανθρωπιστική παρέμβαση με βοήθεια στρατιωτική και άλλες φορές έχουμε πολιτική ανθρωπιστική βοήθεια που δεν θα πρέπει να συγχαίεται με στρατιωτική επιχείρηση. Και γι' αυτό η επικοινωνία είναι ιδιαίτερα σημαντική για να αποφεύγονται παρεξηγήσεις και να αποσαφηνίζουμε τις βασικές αρχές της ανθρωπιστικής δράσης και να ξέρουμε τι άλλες δράσεις μπορεί να βοηθήσουν ε, για την ενίσχυση προστασίας και να στηρίξουν την ανθρωπιστική δράση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον έγκαιρο προγραμματισμό. Στο Τσάντ, όταν στη άλλη αποστολή των Ηνωμένων Εθνών, έγινε ε, επιτόπου ένα έργο ε, ερήμην όμως της κοινωνίας των πολιτών. Δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό και στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, γιατί γνωρίζω ότι οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις χαίρονται ιδιαίτερως που θα ληφθεί υπόψη σοβαρά το θέμα της ασφάλειας. Βέβαια, όσο περισσότερους στρατικούς φορείς έχουμε επιτόπου, τόσο μεγαλύτερα προβλήματα δημιουργούνται για τους ανθρωπιστικούς παράγοντες. Γι' αυτό και είναι σημαντικό να, να στηριζόμαστε σε καλούς αξιωματούχους σύνδεσης για καλύτερο συντονισμό πολιτικού στρατιωτικού σκέλους. Νομίζω ότι η Ότσα έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο εδώ. Ελπίζω να συνεχίσει και στο μέλλον να το κάνει. Και στους μηχανισμούς αυτούς θα πρέπει να δούμε πώς αναμειγνύονται οι ανθρωπιστικοί φορείς. Γιατί στην περίπτωση της Γαλλίας είναι δύσκολο για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις να δίνουν το παρόν στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία ενώ είναι παρούσα γαλλική στρατιωτική δύναμη. Προτιμούν να μένουν στο περιθώριο. Αλλά χρειάζεται ε, απαραίτητη ανταλλαγή πληροφοριών για, την, για τις επιχειρήσεις της ασφάλειας. Οπότε όσο πιο νωρίς μιλάμε και επικοινωνούμε τόσο το καλύτερο. Γι' αυτό και οι μηχανισμοί είναι απαραίτητοι για όταν υπάρχει ταυτόχρονη εμπλοκή και στρατιωτικών και ανθρωπιστικών φορέων. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Ζεράρ τώρα και μετά στο δεύτερο πάνελ. Ευχαριστώ. Αυτό που είπε ο κύριος Γκορένς ε, βρίσκεται στο επίκεντρο και του δικού μας προβληματισμού. Πώς να αποτρέψουμε τις τραγωδίες. Αυτό μας ενδιαφέρει. Και πολύ συχνά οι ανθρωπιστικοί φορείς ακρούν τον κόδωνα του κινδύνου στους πολιτικούς φορείς για τις ανθρώπινες τραγωδίες. Σπάνια έχουμε πολιτικά κινήματα που εξανίστανται ή που αντιλαμβάνουν το πρόβλημα πριν τους ανθρωπιστικούς φορείς, γιατί οι ανθρωπιστικοί φορείς είναι αυτοί που ειδοποιούνται πρώτα απ' όλα από τους τοπικούς πληθυσμούς και είναι αυτό από τις μάρτυρες της κατάστασης. Κύριε Γκέρνς... Είδατε τι έγινε με τη Ρουάντα πριν από μία εικοσαετία και τι συμβαίνει σήμερα με την κεντροαφρικανική δημοκρατία. Πολύ περισσότερο οι φωνές από τον ανθρωπιστικό κλάδο καταδικάζουν τη στρατηγική και επισημαίνουν το πρόβλημα. Πολύ περισσότερο από τις πολιτικές. Η κυρία Γεωργέβα και η κυρία Βαλερία Άμμος... στι αρχέ του Ιουλίου έκρουσαν τον κόδωνα του κινδύνου και ε, χρειάστηκε να περάσει ένα εξάμεινο για να γίνει διάσκεψη. Εδώ και έξι μήνε ε, οι ανθρωπιστικοί φορείς επισημαίνουν το πρόβλημα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Γιατί χρειάστηκε να περιμένουμε τόσο πολύ. Και ίσως το πλεονέκτημα μιας σφαιρική προσέγγισης είναι μια πιο άμεση αντίδραση με τους μηχανισμούς της πολιτικής αντίδρασης, της πολιτικής απόκρισης. Και είναι μια έκκληση και προ του ανθρωπιστικού φορεί μέσω αυτών των προειδοποιήσεων και των συναγερμών να κινητοποιηθούν οι πολιτικοί παράγοντες και να αναλάβουν τις ευθύνες για να αποτρέψουμε, να παρεμποδίσουμε ανθρώπινες τραγωδίες όπως αυτές που συμβαίνουν σήμερα. Οι αντίστοιχες με αυτές της Συρίας που έχουν πολύ πιο πολύ επίπεδη και πολύ σύνθετη δομή. Το έργο των διπλωματών, των κρατών μελών και φορέων όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, οργανώσεων όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι έχουν τις ευθύνες τους και αν ο καθένας αναλάβει την ευθύνη του, θα πρέπει να βρούμε... Καταρχήν, αν ο καθένας έχει την ευθύνη, θα πρέπει να δούμε αν την αναλαμβάνει κιόλα. Εμείς, η κοινότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας, προσπαθούμε να διαπιστώσουμε, να εξακριβώσουμε αν γίνονται σωστά οι διάφορες ε, ενέργειες. Αν ο αποδέκτης ε, λαμβάνει τα κονδύλια που έχουν καθοριστεί για αυτόν. Και θα έπρεπε να έχουμε αντίστοιχου μηχανισμούς για να φέρουμε και τους πολιτικούς πρώτων ευθυνών τους και να εξακριβώσουμε αν έκαναν αυτά που υποσχέθηκαν ή αυτά που όφυλα να κάνουν, ιδιαίτερα σε οξύτατε πολιτικέ κρίσει. Δυστυχώ τέτοιο μηχανισμό για τα πολιτικά θέματα δεν υπάρχει όπω υπάρχει για τα ανθρωπιστικά. Και με αυτή την σφαιρική προσέγγιση, αν καταφέρουμε να προσδιορίσουμε κάποιους συγκριτικούς κανόνες, κάποιους γνώμονες και κριτήρια παρέμβασης ή υλοποίησης ενός πολιτικού προγράμματος, μακάρι να συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα ήμουν ιδιαίτερα ευτυχής. Και τέλος, το θέμα της διαβούλευσης είναι πολύ σημαντικό και ο Κλάου Άρεσεν ο συνάδελφο από το ΕΚΟ, το επισήμανε. Και τα Ηνωμένα Έθνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχουν εμπλακεί σε μια διαδικασία διαβούλευσης. Διαβούλευση όμως δεν σημαίνει κατά ανάγκη ολοκλήρωση, ενσωμάτωση, δεν σημαίνει κατά ανάγκη σφαιρική περιεκτική προσέγγιση. Διαβούλευση λέμε ναι. Γιατί, Γιατί αν μου επιτρέπετε κύριε Ποπόφσκι, δεν θέλουμε οι πολιτικές αποφάσεις να θέτουν σε κίνδυνο τις ανθρωπιστικές δράσεις. Και η συζήτηση που είχαμε για τη Λιβύη ήταν πολύ χρήσιμη, υγιής και απαραίτητη. Γιατί για πρώτη φορά είχαμε ε, κάποιου ευγενική αντιπαράθεση για το πολιτικό και το ανθρωπιστικό πρόγραμμα. Και αυτά ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Και χάρη σε αυτή τη διαδικασία διαβούλευση έγινε αυτή η συζήτηση, όχι στα πλαίσια μια σφαιρική προσέγγιση, συνολική προσέγγιση. Ευχαριστώ. Θα δώσω και πάλι το λόγο στον κύριο Γκιόρε, αλλά παρακαλώ εν συντομή, γιατί έχουμε έξω την Επίτροπο Τζόρτζεβου που περιμένει. Ε, ο κύριος δείχνει ότι όλοι εσείς έχετε πολύ καλή βούληση, οι ομιλητές του πάνελ. Ωστόσο δεν είμαι και τόσο βέβαιος. Δεν έχω πιστεί για τη δυνατότητα αντίδρασής μας σε πολιτικό επίπεδο. Η Ρουάντα δεν έγινε γιατί δεν υπήρχαν μέσα πολιτικά, αλλά γιατί υπήρχε φόβος σε επίπεδο πολιτικό. Ο κύριος Μπούτρος Μπούτρος Γκαλή τα έκανε θάλασσα τότε ε, και ο κύριος Κόφι Ανάν ε, επίσης και οι ευρωπαϊκές χώρες επίσης. Ε, είτε το αγνοήσαμε, είτε είχαμε μια στάση που εκφράζεται καλύτερα με την έκφραση στο κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα. Σε κάθε περίπτωση Υπάρχει πολιτική ευθύνη και δεν είναι ε, το θέμα τα μέσα τα πολιτικά. Μη στρέφουμε τη συζήτηση προς τα εκεί. Ως προς τα μέσα λοιπόν, αυτό το οποίο με εκπλήσει είναι ότι δεν γίνεται αρκετά λόγος για τις αστυνομικές δυνάμεις και την ε, ε, προώθησή τους. Τα περισσότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα σε αυτές τις χώρες είναι, θέματα είναι κυρίως θέματα δημοσίας τάξης. Είναι προβλήματα στο εσωτερικό ε, της κάθε χώρας ή ε, περιοχής και λύνονται με τη δικαιοσύνη αλλά και την αστυνομία. Οι στρατιωτικοί υπάρχουν παντού γιατί δεν υπάρχουν αρκετοί αστυνομικοί. Νομίζω λοιπόν ότι οι αστυνομικές διοκτικές αρχές θα ενοχλούσαν λιγότερο από τις στρατιωτικές αρχές με την παρουσία τους σε μια χώρα. Και από τη στιγμή λοιπόν που στόχος μας είναι να επιλύσουμε εσωτερικές συγκρούσεις, θα πρέπει αυτές οι αρχές ε, ε, να λειτουργούν βάσει των διαταγών των ε, εσωτερικών πολιτικών ευθυνόντων. Νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο κενό από πλευράς μέσων και εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή μας ότι δηλαδή δεν υπάρχει επαρκή ανάπτυξη αστυνομικών δυνάμειων. Από εκεί και πέρα δηλώνω για άλλη μια φορά ότι υπήρξε τεράστια πολιτική αποτυχία στη δεκαετία του 90. Δεν κατάφερε η διεθνής πολιτική να αντιμετωπίσει την ανθρωπιστική κρίση και κυρίως στη Ρουάντα και όχι μόνο. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ επικοδομητική αυτή η συζήτηση. Σας αφήνω όμως σε πολύ καλά χέρια, διότι ο κύριος Νόιζερ θα προεδρεύσει από εδώ και στο εξής. Σας ευχαριστώ και σας χαιρετώ. Okay. Okay. Ε, Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ερχόμαστε τώρα στο δεύτερο μέρος της ακρόασης πριν ε, ξεκινήσουμε με το δεύτερο πάνελ, με μεγάλη χαρά καλωσορίζω την Επίτροπο κυρία Κρυσταλίνα Γεωργίευα, η οποία είναι άρτη αφιχθήσα από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Θα αλλάξουμε λοιπόν λίγο το πρόγραμμα, θα μας ενημερώσει, στη συνέχεια θα έχουμε ερωτήσεις και απαντήσεις της Επιτρόπου και στη συνέχεια θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος της ακρόασης. Καλωσορίσατε κυρία Επίτροπο, έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση αυτή. Σας ευχαριστώ που μου επιτρέπετε να λειτουργήσω ως γέφυρα μεταξύ δύο πάνελ. Το πρώτο ασχολούμενο με την πολιτική και το δεύτερο ασχολούμενο με την εφαρμογή και υλοποίηση. Για να λειτουργήσω λοιπόν καλύτερα ως γεφυροποιός, θα ήθελα να σας δώσω παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζουμε την προσέγγιση μας με βάση τις αρχές μας και γιατί έτσι καταφέρνουμε να κάνουμε τη διαφορά. Ήδη ο Κλάους σας είπε ότι στο πλαίσιο της συνολικής ενιαίας προσέγγισης βρήκαμε μια πολύ καλή λύση για το πώς θα συνδέουμε την ανθρωπιστική βοήθεια με τα υπόλοιπα μέσα ή εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. In but out μέσα μεν αλλά έξω. Αυτός είναι ο ορισμός αυτής της προσέγγισης με τρεις λέξεις και έχει γίνει κατανοητός πλέον από όλους. Και καλό είναι να αναφέρουμε συγκεκριμένα προηγούμενα τα οποία καταδεικνύουν στην πράξη τι σημαίνει να σέβεται κανείς πλήρως τις αρχές της ουδετερότητας, αμεροληψίας και ανεξαρτησίας στο πλαίσιο της ε, πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε συνεργασία με άλλους φορείς ε, από την πολιτική, στρατιωτική σφαίρα ή τη σφαίρα της ανάπτυξης. Ξεκινώ λοιπόν με την εξής υπόθεση εργασίας. Ακριβώς επειδή τηρούμε τις αρχές, μπορούμε με την ανθρωπιστική βοήθεια να συμβάλλουμε στη σταθερότητα, στην ασφάλεια και στην ανάπτυξη χωρίς ε, αυτή τη διάσταση δεν θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε με την ανθρωπιστική βοήθεια. Άλλωστε, βασικός μας στόχος είναι να σώσουμε ανθρώπινες ζωές και να μειώσουμε την οδύνη που υποφέρουν, την οδύνη που έχουν οι άνθρωποι επί τόπου. Και όταν τα καταφέρνουμε, μπορούμε να συμβάλλουμε στην επίτευξη των στόχων των υπολείπων φορέων. Εάν δεν τηρούμε όμως τις αρχές, δεν μπορούμε να συμβάλλουμε θετικά. Θέλω να τονίσω ότι η ανθρωπιστική βοήθεια δεν μπορεί να υποκαταστήσει την εκάστοτε πολιτική λύση που χρειάζεται. Δεν μπορεί να ε, αντισταθμίσει την αποτυχία ε, της πολιτικής. Άρα η ανθρωπιστική βοήθεια δεν μπορεί να επομιστεί ε, τέτοιου είδους στόχους. Εάν όμως εφαρμόζονται σωστά οι πολιτικές, εάν γίνεται σωστή πολιτική με τον τρόπο που θα έπρεπε να γίνεται πολιτική, τότε πράγματι καταφέρνουμε ε, οι άνθρωποι να υποφέρουν λιγότερο. Και φυσικά η μεγαλύτερη κρίση αυτή τη στιγμή είναι στη Συρία πολιτικός ορίζοντας διαγράφεται με πολύ μελανά χρώματα και είναι κάτι που μας απασχολεί ιδιαίτερως από την ανθρωπιστική πλευρά. Στη Συρία γινόμαστε μάρτυρες της αποτυχίας εξέβρεσης πολιτικής λύσης και ως εκ τούτου έχουμε ε, εντελώς αρνητικές ε, συνέπειες και στο ανθρωπιστικό πεδίο. Τις συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα ε, εκφράζονται προσδοκίες για το εξής μπορεί αν αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια στη Συρία και υπάρξει μεγαλύτερη πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια στη Συρία, μπορεί ίσως έτσι να υποβοηθηθεί η πολιτική διαδικασία, να οικοδομηθεί περισσότερη εμπιστοσύνη. Επομένως εμείς σε αυτή την περίπτωση λέμε ξεκάθαρα και φωνάζουμε δυνατά ότι ναι, θέλουμε μεγαλύτερη πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια στην περίπτωση της Συρίας και αν τελικά συμβάλλουμε για περισσότερες πολιτικές διαπραγματεύσει για άνοιγμα, αν θέλετε, πολιτικών διαπραγματεύσεων αυτό είναι καλοδεχούμενο, είναι ευπρόσδεκτο, αλλά δεν θα πρέπει η ανθρωπιστική βοήθεια να είναι όμοιρος των ε, πολιτικών διαδικασιών και τακτικών. Στη Συρία έχουμε λοιμό, έχουμε στέρηση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Αυτό είναι στρατιωτική τακτική που χρησιμοποιείται. Και αυτό είναι λάθος. Επομένως, ε, Πολύ θα μας απασχολήσει η περίπτωση της Συρίας στο μέλλον, όχι μόνο σήμερα, διότι καταδεικνύει την περίπλοκη σχέση μεταξύ της ανθρωπιστικής βοήθειας, της αρχής της ουδετερότητας αμεροληψίας και ανεξαρτησίας από τη μία και της πολιτικής διάστασης από την άλλη, της αποτυχίας δηλαδή της πολιτικής διαδικασίας. Και ελπίζουμε ότι αυτό το τελευταίο θα αντιστραφεί, δηλαδή η πορεία αποτυχίας θα ανακοπεί. Όλα αυτά τα χρόνια που είμαι επίτροπος, έχω δει πώς εφαρμόζεται στην πράξη αυτή η αρχή και όλες αυτές οι αρχές και πόσο μεγάλη αξία έχουν όταν εφαρμόζονται. Και θα δώσω παραδείγματα τα οποία με καθιστούν ε, μεγάλη υπέρμαχο της ε, κυριαρχής προσέγγισης στην ανθρωπιστική βοήθεια και ε, ο βασικός λόγος είναι ο εξής. Μία από τις πρώτες μου εμπειρίες ήταν στην Ιεμένη. Εκεί Ακριβώς χάρη στην αρχή της ουδετερότητας αμεροληψίας και ανεξαρτησίας καταφέραμε να διαπραγματευτούμε με τον ΙΠΑ το εκπρόσωπο κύριο Γκουτιέρες έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση η λειτουργή της ανθρωπιστικής βοήθειας στο βόρειο μέρος ε, της ε, χώρας σε ε, περιοχές όπου έλεγχαν οι Χούτι. Και εάν δεν το είχαμε καταφέρει αυτό, τότε ούτε η κυβέρνηση θα το είχε επιτρέψει, ούτε οι ίδιοι οι Χούτι θα είχαν δεχθεί να τους επισκεφθούμε. Όμως τα καταφέραμε διότι το επιχείρημά μας ήταν ακριβώς αυτό, το ανθρωπιστικό σκέλος, ότι θέλουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους εκεί. Μας επέτρεψαν λοιπόν να δούμε τους ε, ε, επικεφαλείς τους, ε, των Χούτι. Συζητήσαμε με αυτούς και επιτράπηκε η πρόσβαση στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού. Και 300.000 άνθρωποι υποφελήθηκαν από αυτή τη βοήθεια. Για κάποιους ήταν θέμα ζωής και θανάτου. Και αυτό δείχνει πόσο μεγάλη αξία έχουν αυτές οι τρεις αρχές. Αλλά και στην Κυργυζία, όπου θα θυμάστε ότι υπήρξε μια τεράστια εθνοτική σύγκρουση μεταξύ Κυργίζεων και Ουσμπέκων, που εθνοτική ομάδα Ουσπέκων, ε, κάτι το οποίο οδήγησε ε, σε 250.000 εκτοπισμένους στο Ουσμπέκισταν μέσα σε λίγες ε, μέρες. Έσκαψαν μία τρύπα στα σύνορα βάθους τριών μέτρων και για να τα περάσουν. Και όσοι έμειναν εκεί και στις ε, γύρω περιοχές μου είπαν επανειλημμένως είμαστε ευγνώμονες για την οικονομική σας στήριξη αλλά είμαστε περισσότερο από όλα ευγνώμονες διότι χάρη σε αυτή τη στήριξη έχουμε εδώ ανθρώπους με τη σακάκια, ε, με τα ε, σήματα του Ερυθρού Σταυρού και άλλων ε, διεθνών οργανώσεων και αυτοί εκφράζουν τις ελπίδες μας για σταθερότητα ενώ ε, οι σφαίρες ε, πέφτουν γύρω μας με πολύ μεγάλο ρυθμό, πολύ έντονο ρυθμό. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι αυτή η αρχή της αμεροληψίας, ουδετερότητας και ανεξαρτησίας είναι που έκανε τη διαφορά. Είναι αυτή που σταμάτησε κάποιες από αυτές τις σφαίρες που πετούσαν στον αέρα. Και Χαίρομαι διότι οι εταίροι μας με την παρουσία τους εκεί συνέβαλαν στην ασφάλεια ε, χιλιάδων, δεκάδων χιλιάδων και περισσότερων μάλιστα ανθρώπων. Πιστεύω ακραδάντως από τις εμπειρίες που είχα και στο Μαλί και στην ακτή του Ελεφαντοστού και στην κεντροαφρικανική δημοκρατία ότι η ανθρωπιστική κοινότητα ακριβώς χάρη ε, στην υψηλότερη ανεκτικότητα, αν θέλετε, που έχει στην ανασφάλεια, επειδή βασίζεται σε αυτή την αμεροληψία, την ανεξαρτησία και την ουδετερότητα, μπορεί να παραμείνει σε περιοχές όπου βεβαίως δεν μπορεί να λάβει χώρα καμνενός είδου, ε, είδους ανάπτυξη προς το παρόν. Μιλώ για το Βόρειο Μαλί ή για τις ε, περιοχές της ακτής του Ελεφαντοστού όπου έχουμε τις συγκρούσεις, αλλά και ε, αυτή τη στιγμή στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Επειδή λοιπόν έχουμε τους λειτουργούς της ανθρωπιστικής βοήθειας επιτόπου, τους αφήνουν να κάνουν τη δουλειά τους άνθρωποι εξαιρετικά κακοί, οι εξτρεμιστές για παράδειγμα στο Βόρειο Μαλί. Αφήνουν την ανθρωπιστική δράση να λειτουργεί όσο καλύτερα μπορεί. Οι μαχητέ Ελέκα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, όσο κακή και αν είναι, επιτρέπουν στην ανθρωπιστική βοήθεια να εφαρμοστεί. Και... Έτσι, έχουμε την υψηλή ανεκτικότητα απέναντι στον κίνδυνο και έτσι μπορούμε να παράσχουμε τις στοιχειώδεις υπηρεσίες και να έχουμε επιχειρήσεις αποκατάστασης και 23 ε, εκατομμύρια για παράδειγμα στο Μαλί για επαναφορά των βασικών υπηρεσιών, ηλεκτρισμό, ίδρυυση, υγειονομικές υπηρεσίες, εκπαίδευση. Έτσι δημιουργείται πρόσφορο κλίμα για επιστροφή του κόσμου. Και όταν επιστρεφθούν οι εκτοπισμένοι θα ε, αποκατασταθούν και οι διοικητικοί θεσμοί και θα επανέλθει στην ομαλότητα το Βόρειο Μπαλί. Και στην ακτή του Ελεφαντοστού. Εκεί δημιουργήσαμε την εταιρική σχέση για τη μετάβαση και περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ με βάση την παρουσία ανθρωπιστικών οργανώσεων προσπαθήσαμε να παράσχουμε στοιχειώδεις υπηρεσίες και να συμβάλλουμε στην επαναφορά της ομαλότητας και στην ε, επαναφορά των κρατικών θεσμών. Και πολύ συχνά στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία έχουμε ακούσει για τις επιτυχίες, επιτυχίες μας ε, παρεμβάσεις. Και η σημερινή μέρα για μένα και το επιτελείο μου είναι μια λαμπρή μέρα, γιατί έχουμε καταφέρει να μην μείνει πια λησμονημένη η κεντροαφρικανική δημοκρατία. Έχουμε 100 εκατομμύρια σε αναλήψεις υποχρεώσεων και έτσι θα έχουμε συνεργασία του αναπτυξιακού σκέλους με το ανθρωπιστικό για να συμβάλλουμε με βάση τις αρχές μας να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Έχω ξεπεράσει το χρόνο μου και σας ζητώ συγγνώμη. Ξεπέρασα κατά 1,5 σχεδόν λεπτό το χρόνο που μου δώσατε, αλλά πιστεύω ότι με τα παραδείγματα αυτά θα δημιουργήσουμε τη γέφυρα από, την, από τα λόγια στα έργα, από, το, από τη χάραξη της πολιτικής στην εφαρμογή της. Σας ευχαριστούμε κυρία Γκιαόργεβα, κυρία Επιτρόπη. ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η ομιλία σας και όπως είπατε και στις τελευταίες σας φράσεις, είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί επιτέλους ε, το θέμα της κεντροαφρικανικής δημοκρατίας ε, μπαίνει στο προσκήνιο και μαζί με τη Συρία είναι από τα πιο σημαντικά θέματα και χαίρομαι που ξαναβρίσκονται στο επίκεντρο. Ο κύριος Κορτές Λάστρα, η κυρία Κρές και μετά ο κύριος Γκέρενς. Κύριε Κορτές Λάστρα, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Πριν είχαμε διαφορετική σύνθεση του πάνελ, και είχα την αίσθηση ότι σε πολλές περιπτώσεις μας λείπει η πολιτική συμφωνία ώστε να μπορέσουμε από κοινού με ανθρωπιστικές επιχειρήσεις και δράσεις να έχουμε πολύ πιο θεαματικά αποτελέσματα από αυτά που έχουμε μόνο μέσω της αμυγούς ανθρωπιστικής μας βοήθειας. Θα ήθελα ευκαιρία, να σας ευχαριστήσω μεν για την παρουσία σας και να σας κάνω και μία ερώτηση. Γιατί ακούσαμε τελευταία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και έχουμε και την αίσθηση αυτή στην Επιτροπή μας ότι κάθε μέρα που περνά έχουμε όλο και περισσότερα θέματα επιτάπητος σε σχέση με την ανθρωπιστική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακούσαμε όμως και διαβάσαμε ότι η κατάσταση του ΕΚΟ, του Τμήματος Ανθρωπιστικής Βοήθειας, έχει οικονομικά προβλήματα, αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Οπότε εμείς ε, Θεώρησαμε ανέκαθεν την ανθρωπιστική βοήθεια ως προτεραιότητα και της δικής μας Επιτροπή. Και γι' αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω. Αυτή τη στιγμή, πού έγινε το πρόβλημα, στις κυβερνήσεις, γιατί μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα. Θα θέλαμε η σύσσωμη επιτροπή μας να βοηθήσει στο να απεμπλακεί κατάσταση ώστε να συνεχίσει να αρέει η ανθρωπιστική βοήθεια όπως γινόταν μέχρι τώρα. Γιατί έχουμε πολλές καταστάσεις κρίσεως που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και θα ήθελα απάντηση. Ευχαριστώ κυρία Κρέσ. Ευχαριστώ. Αναφερθήκατε στο θέμα της κεντροαφρικανικής δημοκρατίας. Όντως είναι επίκαιρο το θέμα και με ενδιαφέρει και ιδιαίτερος για τη Μεγαλίδα όπως αντιλαμβάνεστε. Είπατε ότι σήμερα για σας η μέρα ήταν πολύ σημαντική, γιατί βρέθηκε στο επίκεντρο αυτό το θέμα. Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες, τι ακριβώς δηλαδή θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Σας ευχαριστώ και κυρίως για τα σύντομη ερώτησή σας. Ο κύριος Γκέρενς, σας ευχαριστώ. Η, δυστυχώς η δική μου ερώτηση θα είναι πιο μακροσκελής. Την περασμένη εβδομάδα Ε, είχαμε επαφές με κάποιους εκπροσώπους των ανθρωπιστικών οργανώσεων που φοβόνταν ότι θα είχαμε δραστικές περικοπές ε, του προϋπολογισμού για τα ανθρωπιστικά θέματα. Η ερώτηση μου είναι απλούστατη λοιπόν. Αντιμετωπίζετε προβλήματα στον προϋπολογισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ε, βλέπω ότι νεύεται καταφατικά. Uh, uh ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Να ξεκινήσω και να απαντήσω μαζί στις ερωτήσει του κ. Κόρτη και του κ. Γκόρεντ, γιατί συνδέονται με το ίδιο θέμα. Τι αντιμετωπίζουμε. Πρόβλημα ροής ε, χρημάτων. Θα εκπληρώσουμε όλες μας τις δεσμεύσεις. Εκφράστηκε στις αρχές της ε, προηγούμενης εβδομάδας ε, μία ανησυχία ότι ενδεχομένως να μην είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε όλες μας τις δεσμεύσεις ε, βάσει της απόφασης που είχαμε λάβει για να συνδράμουμε στα άτομα που αντιμετωπίζουν καταστάσεις κρίσης σε όλο τον κόσμο. Θα εκπληρώσουμε λοιπόν τις αποφάσεις μας το έπακρον. Αλλά έχουμε ένα θέμα σε ό,τι αφορά την διαχείριση της ροής χρημάτων. Οι χρηματοποιητικές αρχές μας βοηθούν να επιλύσουμε το θέμα αυτό. Και γιατί αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα αυτό. Γιατί πολύ απλά πέρσι η χρονιά ήταν εξαιρετική. Είχαμε πολύ πιο πολλά να κάνουμε τελικά από τον αρχικό μας προϋπολογισμό. Στο τέλος είχαμε χορηγήσει 1.353 εκατομμύρια ευρώ σε ανθρωπιστική βοήθεια. Επιπλέον κινητοποιήθηκαν και άλλα τμήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρίως για την κρίση στη Συρία, για να συνδράμουν τις σχετικές κοινότητες, το Λίβανο, την Ιορδανία. Για να σας δώσω ε, μια ένα παράδειγμα για το πόσο δραματικό ήταν το έτος. Ήμουν στο Κουβέιτ την προηγούμενη εβδομάδα για το δεύτερο συνεδρίο σε ό,τι αφορά τους δωρητές και καταμετρήσαμε το τι έχει χορηγήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην, στο λαό της Συρίας από την προηγούμενη συνεδρίο. 136 εκατομμύρια ευρώ, δολάριο είχαμε δεσμευτεί να δώσουμε στην πρώτη συνεδρία ε, του Κουβέιτ, το επταπλάσιο, ένα δισεκατομμύριο δολάρια τελικά χορηγήσαμε και για την Ιορδανία και για τη Λιβύα. Μια έκτακτη κατάσταση η οποία απαιτεί έκτακτα μέτρα. Και από πάνω είχαμε την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, τον Νότιο Σουδάν, τις Φιλιππίνες. Υπό το νέο λοιπόν καθεστώς χρηματοδότησης, όπως ξέρετε, οι πιστώσεις πληρωμών ε, βρίσκονται υπό πολύ αυστηρή διαχείριση. Και αυτό γιατί μας δημιουργεί πρόβλημα. Οι δεσμεύσει εφαρμόζονται άμεσα, εντό μηνών και εντό ενό έτους το αργότερο, όταν οι δεσμεύσει είναι πιο υψηλέ από τι πιστώσεις πληρωμών, αντιμετωπίζουμε πρόβλημα. Και πώ το επιλύουμε, δύο πράγματα κάνουμε. Αφενός, αναθεωρήσαμε όλες μας τις δραστηριότητες για να εξασφαλίσουμε ότι οι προτεραιότητες μας χρηματοδοτούνται άμεσα και κατά προτεραιότητα και αυτές οι οποίες ε, ε, όπου υπάρχει περιθώριο αργότερης ε, εφαρμογής μετατίθενται προκειμένου να λάβουμε πιο πολλές πληρωμές πιστώσεων πιο πολλές πιστώσεις πληρωμών αργότερα το χρόνο. Η χρηματοδοτική αρχή λοιπόν, η αρχή προϋπολογισμού εξετάζει κατά πόσον υπάρχει ανάγκη μετακίνηση σε άλλο πρόγραμμα προκειμένου να ενισχυθούν οι πιστώσεις πληρωμών. Όπου μπορούν να το κάνουν, το κάνουν αυτό. Συνολικά έχω την αίσθηση ότι και είμαι αισιόδοξη ότι θα τα καταφέρουμε σε βάθος χρόνου, σε όλο το έτος. Αλλά θα πρέπει να επιλύσουμε αυτό το συστημικό πρόβλημα για την ανθρωπιστική βοήθεια σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις και τις πιστώσεις ε, πληρωμών που δεν ε, συμμορφώνονται, που δεν είναι αντίστοιχες. Γιατί δάλλως αντιμετωπίζουμε πρόβλημα εφαρμογής μακροπρόθεσμα. Γιατί για παράδειγμα ένας δρόμος παίρνει χρόνια μέχρι να κατασκευαστεί και ε, έτσι, για παράδειγμα, δεν μπορεί κανείς να αγοράσει φάρμακα με μια υπόσχεση, μόνο με χρήμα, με ρευστό μπορεί κανείς να αγοράσει φάρμακα. Και έχουμε συνεργαστεί πολύ στενά με τους εταίρους μας για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό, να το κατανοήσουμε και να το λύσουμε. Και ε, επίσης ελπίζω να μπορέσουμε να συνεργαστούμε και με εσάς για να επιλύσουμε αυτό το συστημικό πρόβλημα προκειμένου να μην ανακύπτει διαρκώς στο μέλλον. Γιατί δεν πρόκειται να αποτελέσει αυτό το έτος ένα τόσο εξαιρετικό έτος, τόσο έκτακτο σε ανάγκες. Αλλά το γεγονός είναι ότι μπορεί να υπάρξουν ε, παράλληλες κρίσεις, οι οποίες θα πλήξουν παράλληλα. Αυτός ο κίνδυνος είναι πολύ πραγματικός. Είναι μεγάλος, ιδιαίτερα και εν ώψη του ευάρτου κλίματος. Υποβάλαμε μία πρόταση για ένα αποθεματικό για τις πιστώσεις αυτές να είναι πιο, πολύ, πιο πολλές και από το μαθηματικό. Αλλά η πρόταση αυτή δεν έτυχε υποστήριξη. Και από εκεί πηγάζει και το πρόβλημα ρευστότητας. Αν σας ενδιέφερε, εμείς Θέλουμε να επιλύσουμε αυτό το συστημικό ζήτημα. Το έχω συζητήσει και με διάφορα κρατημέλη. Και υπάρχει ασφαλώς μια γενική κατανόηση για το θέμα αυτό εν ώψη και των όσων συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Αλλά αυτό θα πρέπει να μεταφραστεί σε μια συστημική λύση του θέματος. Για να μην αντιμετωπίζουμε διαρκώς το ίδιο θέμα. Κατά μία έννοια λοιπόν κύριε Γκούρεντς έχουμε βρει μία λύση, αλλά δεν πρόκειται για μία αέναη λύση. Θα πρέπει να επιλύσουμε το πρόβλημα και να το χτυπήσουμε στη ρίζη της. Στην ανθρωπιστική βοήθεια θα πρέπει να είναι αντίστοιχες οι δεσμεύσεις και οι πιστώσεις, πολύ απλά λόγω της φύσεως της εργασίας μας, της δουλειάς μας. Για το δεύτερο ερώτημα για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Σήμερα έχουν συμβεί τρία θετικά πράγματα για το λαό που υποφέρει. Καταρχάς η απόφαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων να υποστηρίξει τις ε, συνεισφορέ των κρατών μελών σε ό,τι αφορά την ασφάλεια στην κεντροαφρικανική δημοκρατία. Αυτό θα αναπτυχθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια, αλλά τι σημαίνει αυτό επί τη αρχή, ότι οι Ευρωπαίοι θα συνδράμουν την Γαλλία και τη Μίσκα με στρατεύματα, με εξοπλισμό και με άλλου στρατιωτικό εξοπλισμό. Εμεί, από πλευρά ανθρωπιστική κοινότητα, ε, το καλωσορίζουμε αυτό. Σπάνια αναφέρουμε ε, ότι υποστηρίζουμε τέτοια ε, στρατιωτική παρέμβαση, αλλά είναι πραγματικά τραγική η κατάσταση. Πυρπολείται ο κόσμος, ακροτηριάζονται με μαντσέτες. Οι δε θρησκευτικέ σειράξει έχουν ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Θα πρέπει λοιπόν να το ελέγξουμε αυτό. Δεύτερη θετική εξέλιξη. Νέο πρόεδρο. Νέο μεταβατικό πρόεδρο εκλέχθη. Μάλλον, συγγνώμη, νέα μεταβατική πρόεδρος. Γυναίκα, γυναίκα. Και με τον σεβασμό που τρέφω σε όλους τους άντρες, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι πάρα πολύ καλή αυτή η είδηση, γιατί τίνουμε οι γυναίκες να έχουμε μία ηρεμία πνεύματος. Ελπίζουμε λοιπόν αυτό να βοηθήσει. Είναι και αντίμερχος στην Παγκή. Αυτό σημαίνει ότι ελπίζουμε ότι θα έχει και κάποια διοικητική εμπειρία. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι όλα αυτά ασφαλώς θα υλοποιηθούν, ότι αποτελούν όντω καλέ ειδήσει, είναι εν πάση περιπτώσει όμω τουλάχιστον ενθαρρυντικά. Υποστηρίχθηκε εκτενώ στο δεύτερο γύρο των εκλογών. Ελπίζουμε να είναι ισχυρή η εντολή τη Και τρίτη είδηση θετική είναι ότι η συνδιάσκεψη, η ανθρωπιστική που έλαβε χώρα σήμερα το πρωί, συμπεριέλαβε 45 χώρε, όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετείχαν, 18 κράτη-μέλη συμβάλλουν, συνεισφέρουν οικονομικά από Ιαπωνία, από, την, από τη ΣΥΠΑ, μεγάλες συνεισφορές και από τον Καναδά. 35 διεθνείς οργανώσεις ε, συμμετείχαν, μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ο ΙΕ, η Διεθνής Τράπεζα, η Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης, ε, μεγάλες δεσμεύσεις και από αυτές τις οργανώσεις για μέτρα σταθεροποίησης της χρηματοδότησης και καταλήξαμε σε εκπληκτικά υψηλό ποσό σε σχέση με αυτά που λάμβανε ε, στο παρελθόν η κεντροαφρικανική δημοκρατία 500 εκατομμύρια μέτρα σταθεροποίησης αμυγός ανθρωπιστικής φύσεως. Ακριβώς αυτό θα πρέπει να κάνουμε, σταθεροποίηση μέσω της καλύτερης επίδειξης της συνολικής αυτής προσέγγισης, με σεβασμό των αρχών που αναφέραμε προλίγου. Αυτό έγινε σήμερα. Ελπίζουμε η 20 Ιανουαρίου να μείνει στην ιστορία ως σημείο καμπής για την κεντροαφρικανική δημοκρατία. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίτροπε, νομίζω ότι ήταν πραγματικά απαραίτητο να σας αφιερώσουμε τα πέντε λεπτά παραπάνω. Ε, κύριε Γκέρονς, δεν έχουμε δυστυχώς χρόνο. Ευχαριστώ. Θέλω να θέσω ένα σημαντικό ερώτημα. Είπατε ότι το 2013 ήταν μια εξαιρετική χρονιά. Ούτε το 2014 θα ήταν συνηθισμένη χρονιά. Αυτό δείχνουν οι ενδείξεις. Στα συστημικά προβλήματα στα οποία αναφερθήκατε, επανειλημμένος προσφύγατε σε διάφορες ε, πρακτικές που προσπαθούν να επιλύσουν τα προβλήματα σε βραχυπρόθεσμη βάση και είπατε ότι κανείς δεν αγοράζει φάρμακα με τις υποσχέσεις που του δίνονται. Ζητώ λοιπόν ένα και ρωτώ το εξή. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στο Ευρωπαϊκό Αρχιτεκτόνημα. Δεν μπορεί να προκαταβάλει τα απαραίτητα κονδύλια επί τη βάση της υπόσχεσης εκεί όπου λείπουν τα φάρμακα και όπου η άλλη επιλογή είναι απλά να αφήσουμε τον κόσμο να πεθαίνει. Θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Επομένως, αν υπάρχει υπόσχεση που θα έχει αναλυφθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε δίνεται εμπιστοσύνη, νιώθει εμπιστοσύνη μια τράπεζα να δώσει αυτή την προκαταβολή και έτσι μπορούμε να, κάνουμε την προσέγγιση. Να την κάνουμε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να προσεγγίσει περισσότερο ε, αυτές τις περιοχές. Και νομίζω ότι με το δικό σας κύρος θα μπορείτε να την πείσετε. Απάντηση της Επιτρόπου. Προς το παρόν θεωρούμε ότι οι μεταφορές μεταξύ ε, των υποκλάδων του, της επικεφαλίδας 4 ε, είναι αρκετές και δεν θα χρειαστεί. Σωστή όμως η παρατήρησή σας. Όταν οι συνθήκες είναι εξαιρετικές θα πρέπει να είμαστε πιο επινοητικοί, πιο δημιουργικοί για να κινητοποιήσουμε επιπρόσθετα κονδύλια και για την ασφάλεια των πολιτών μας. Γιατί αυτά τα οποία κάνουμε για να σταθεροποιήσουμε το Λίβανο και την Ιορδανία μεταφράζονται σε μείωση του κινδύνου για εσάς, για εμάς, για τους πολίτες μας η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ομολογώ ότι δεν το είχα σκεφτεί. Θα το σκεφτώ, θα μιλήσω με τον διοικητή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, τον κύριο Χόγερ, σίγουρα. Ωστόσο αυτό το οποίο έχουμε εξετάσει είναι το εξή. Κάποια από τα κονδύλια που δίνουμε για τον ανταγωνισμό, μήπως θα μπορούσαμε να τα αξιοποιήσουμε για να έχουμε επιπρόσθετα έσοδα για ανθρωπιστική βοήθεια. Είναι χρήματα τα οποία δεν περιμένουν να πάρουν πίσω τα ε, κράτη-μέλη είναι χρήματα τα οποία επιστρέφονται στα κράτη-μέλη. Εάν θέλουν όμως τα κράτη-μέλη να προστατεύσουν τα συλλογικά συμφέροντα της Ευρώπης σε περίπτωση μιας κρίσης τόσο πρωτοφανούς όπως είναι η κρίση, τότε μπορούν να αποφασίσουν ότι θα παρετηθούν από το να λάβουν τα χρήματα και να τα εκχωρήσουν στην ανθρωπιστική βοήθεια και άρα θα σφυριλατηθεί, θα ενισχυθεί η ανθρωπιστική δράση. Αλλά βεβαίως αυτό είναι επιλογή των κρατών μελών και θα πρέπει να δούμε ε, κατά πόσο ανοίγεται εκεί ένας δρόμος ή όχι. Προσπαθώ όμως να σκεφτώ πιο επινοητικά, πιο δημιουργικά και λέω ότι Πρέπει να βρούμε τρόπους να γεννήσουμε εντό εισαγωγικών χρήμα χωρίς να πλήττουμε τη δημοσιονομική πειθαρχία και χωρίς να αυξάνουμε τη δημοσιονομική πίεση στα κράτη-μέλη. Συλλέγουμε 1,7 δις ευρώ από τις ε, ε, τράπεζες. Ένα ε, ελάχιστο ε, κομματάκι από αυτά τα χρήματα ε, να είχαμε θα διανύαμε τεράστια απόσταση στο δρόμο της ανθρωπιστικής βοήθειας. Αλλά βεβαίως θα έρθω σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να δω πώς μπορούμε να συνεργαστούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Γκέρενς γιατί πραγματικά η ιδέα σας είναι καταπληκτική. Βέβαια. η Επιτροπή μας να στηρίζει την Επίτροπο Γεωργίευα και ελπίζω να έχουμε καλές και σαφείς απαντήσεις και αντιδράσεις για την κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και κάποιες ιδέες για να βρούμε και νέα έκτακτα κονδύλια για την ανθρωπιστική βοήθεια. Σας ευχαριστούμε θερμά που ήρθατε. Ξέρουμε ότι είναι πολύ φορτωμένο το πρόγραμμά σας και σας ευχαριστούμε θερμά για το έργο σας. Ευχαριστώ και περνάμε τώρα στο δεύτερο πάνελ μας. Να καλέσω παρακαλώ τους καλεσμένους μας από το δεύτερο πάνελ. Συγγνώμη για την πίεση χρόνου, ελπίζω να τα καταφέρουμε στα τρία τέταρτα που μας έχουν απομείνει.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 six Καλώς ήρθατε στο δεύτερο πάνελ της ακροασής μας. Να σας παρουσιάσω τον κύριο Τζιλς Χάσολ, τον κύριο Ζαν Φιλίπ Γκανάσια, το λέω σωστά. Και λυπάμαι που σας αναφέρω τελευταία την κυρία Σελήνη Μίας. Μου λέει ο σύμβουλός μου ότι έχετε ένα 7 λεπτό καθένας. Ελπίζω να σας ε, αρκέσει. Ο κύριος Χάνσουλ, σας ευχαριστώ και ευχαριστώ που καλέσατε την Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, την ICRC, για να σας μιλήσει για αυτό το πρόβλημα της σύγχυσης ε, που υπάρχει. Και θα μιλήσω κυρίως ε, για τις ε, περιοχές όπου έχουμε ένοπλες συγκρούσεις. Ο Ερυθρός Σταυρός έχει κυρίως δράσεις προστασίας άμαχο πληθυσμού, προστασία τραυματιών, κρατουμένων, καθώς και κάποιες επιχειρήσεις συνδρομής, παροχής βοήθειας η στρατηγική, καταρχήν ποια είναι η στρατηγική του Εθνικού, του, της Διεθνής Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού για να φτάσει στους ε, αναξιοπαθείς. Αναφέρθηκαν ε, οι βασικές αρχές ε, στην απογευματινή συζήτηση που είχατε. Καταρχήν, αμεροληψία, ανεξαρτησία και ουδετερότητα. Αυτές είναι οι τρεις βασικές αρχές. Μπορεί να ακούγεται κάπως θεωρητικό αυτό, αλλά όπου και αν δραστηριοποιούμαστε πάντα εφαρμόζουμε την ίδια συνταγή. Να φτάσουμε κοντά στο, στο τοπικό πληθυσμό και να εφαρμόσουμε κυρίως ε, δράσεις που στηρίζονται σε ουδετερότητα και ανεξαρτησία. Έτσι θα κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των ε, πληθυσμών και των διαφόρων πλευρών της ε, σύγκρουσης και αυτή η εμπιστοσύνη θα κάνει το έργο μας πιο εύκολα αποδεκτό και θα έχουμε καλύτερη πρόσβαση στον πληθυσμό. Το πρόβλημα υπάρχει όταν δημιουργείται μια σύγχυση, γιατί έτσι μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο ολόκληρη η στρατηγική μας. Το θέμα της σύγχυσης θα ήθελα να το παρουσιάσω δίνοντας παραδείγματα από τρεις διαφορετικές καταστάσεις. Δεν λέω ότι θα είναι εξαντλητικά αυτά τα παραδείγματα και θα καλύψουν όλες τις ε, πιθανές περιπτώσεις. Θα περιοριστώ όμως σε τρία παραδείγματα. Καταρχήν, μερικές φορές η ανθρωπιστική βοήθεια μπορεί να θεωρηθεί ως εργαλείο για άλλους ε, στόχους, είτε στρατιωτικούς, είτε ευρύτερους πολιτικούς στόχους. Όταν υπάρχει τέτοια αντίληψη, υπάρχει κίνδυνος για τις ανθρωπιστικές οργανώσεις όπως ε, τον Ερυθρό Σταυρό να μην γίνουν αποδεκτές ε, στο θέατρο των επιχειρήσεων, κάτι που θα ε, φέρει σε κίνδυνο το προσωπικό μας, είτε είναι τοπική είτε είναι αποσπασμένη και θα δημιουργήσει κίνδυνο και θα υπονομεύσει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον πληθυσμό που τη χρειάζεται. Επίσης, όταν έχω μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ή περιεκτική προσέγγιση, εκεί που δηλαδή ο στρατητικός ε, παράγοντας θέλει να βοηθήσει την, τις δικές μας δράσεις, στην περίπτωση του Αφγανιστάν, για παράδειγμα, είχαμε τέτοια περίπτωση, εκεί είχαμε κάποιες ε, επαρχιακές ε, ομάδες για την ανασυγκρότηση. Περισσότερες τώρα έχουν κλείσει, έχουν ολοκληρώσει τα προγράμματά τους, αλλά ήταν χαρακτηριστικό παράδειγμα, χαρακτηριστική περίπτωση που έχουμε ένα στρατιωτικό σκέλος, ένα πολιτικό σκέλος και έχουμε και τεχνοκράτες ε, ε, ή μάλλον τεχνικό προσωπικό, μπορεί να είναι μηχανική, πολιτική μηχανική, γιατρή, ιατρικό προσωπικό. Οπότε θέλουμε εκεί να επεκτείνουμε την εξουσία της κεντρικής αρχής της επαρχίας. Και αυτό που είδαμε στην πράξη είναι ότι έχουμε αυτούς τους ε, μηχανικούς του PRT των επαρχιών αυτών που ηγούνται προγραμμάτων ίδρευσης για τις τοπικές κοινότητες ή έχουμε ιατρικό προσωπικό που, πηγαίνει σε απομονωμένες περιοχές για να παρέσει ε, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αλλά υπάρχει πρόβλημα με την επικάλυψη κάποιων αμυγός ανθρωπιστικών προγραμμάτων ή προγραμμάτων που εφαρμόζονται από ανθρωπιστικέ οργανώσει και στρατιωτικών προγραμμάτων. Τότε δημιουργείται σύγχυση στα μάτια του τοπικού πληθυσμού και αυτό μας απασχολεί και μας προβληματίζει. Έχουμε και ένα δεύτερο είδος ε, ολοκληρωμένη προσέγγισης, όπου έχουμε τις ε, ολοκληρωμένε αποστολέ ε, του ΟΗΕ. Εκεί έχουμε μερικέ αποστολέ όπου έμειναν στο περιθώριο ανθρωπιστικές οργανώσεις, αλλά το θέμα το πώς μας αντιλαμβάνονται είναι βασικό στοιχείο. Στην περίπτωση του Μαλή, για παράδειγμα, οι συνάδελφοί μου φοβούνται ότι η μήνεσμα έχει ισχυρή εντολή ασφάλειας και σκοπεύει να δρομολογήσει κάποια προβλήματα άμεσου αντικτύπου. Υδροδότηση, για παράδειγμα, πρόγραμμα και εκεί υπάρχει αυτή η επικάλυψη που δημιουργεί σύγχυση. Ένα τρίτο σύντομο παράδειγμα, κάπως διαφορετικό από την ασφαιρική ολοκληρωμένη προσέγγιση, εκεί που οι ανθρωπιστικές οργανώσεις συμμετέχουν στη δημιουργία υποδομών, όπως στη Σομαλία. Εκεί ο Ερθρός Σταυρός πρόσφερε μια προστιθέμενη αξία συμμετέχοντας σε προγράμματα δημιουργίας θεσμικών δομών, υποδομών, στη Γεωργία, στην υγεία, στην υδροδότηση, αλλά είναι πολύ λεπτή η γραμμή ε, που λαμβάνει υπόψη ο Ερθρός Σταυρός, γιατί μερικές φορές εργάζεται σε ε, περιοχές που ελέγχονται από την άλλη πλευρά. Οπότε η σωστή, ο σωστός διαχωρισμός και η σωστή αντίληψη είναι θέμα ζωής και θανάτου μερικές φορές και θα πρέπει να γίνεται αυστηρός έλεγχος. Ένα λεπτό μου έμεινε να μιλήσω για τα μαθήματα που έχουμε διδαχθεί, για τα συμπεράσματα που έχουμε αντιλήσει. Δεν υπάρχουν και πολλά καινούργια στοιχεία εδώ. Η πρώτη μου αντίδραση ήταν ότι η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού θα κρατούσε αποστάσεις από βασικές στρατητικές και πολιτικές επιχειρήσεις επιτόπου, ταυτόχρονα θα έχει διμερή διάλογο με τις ανεχόμενες πλευρές. Καταρχήν για να εφαρμόσει την εντολή της και, την, και να δώσει στις ενεχόμενες πλευρές να καταλάβουν την εντολή και τις, τους περιορισμούς αυτής της προσέγγισης και να αποσαφηνίσει ότι δεν ε, συμμετέχει σε κανένας είδους σφαιρική ολοκληρωμένη προσέγγιση. Επίσης, ε, συνειδητοποίησαμε την ανάγκη σωστών μηχανισμών συντονισμού και συμμετέχουμε σε αυτούς ε, με σεβασμό της εντολής μας, μερικές φορές ακόμη και ως παρατηρητές. Πάντως είναι πολύ σημαντικό επιτόπου να έχουμε τέτοιο καλό συντονισμό για να αποφευχθούν τα προβλήματα. Και τέλος, να πω ότι διαπιστώσαμε ότι η κατάρτιση του πολιτικού και στρατιωτικού προσωπικού που αναπτύσσεται επιτόπου για τα ανθρωπιστικά θέματα είναι πολύ σημαντικός παράγοντας, θα έλεγα ναυραλγικός, για να βελτιώσουμε την αμοιβαία κατανόηση και τον αμοιβαίο σεβασμό των εντολών μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Πολύ συγκεκριμένα και σαφή τα παραδείγματα που μας δώσατε. Να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Γκανάσια που έχει πλούσια πείρα από το Τζάτ, το Κονγκό, την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και ούτω καθεξής. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε ως πρώην στρατιωτικό για να μιλήσω για αυτό το θέμα ε, με το οποίο έχει ασχοληθεί και στο Τσάντ αλλά και τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Η σχέση του πολιτικού με το στρατιωτικού σκέλος, λοιπόν, πώς ορίζεται η ένταση που συχνά υπάρχει ανάμεσα σε αυτούς τους δύο διαφορετικούς κόσμους θα έλεγα. Ε, θα έλεγα ότι επί τόπου αυτή τη σχέση ε, την ορίζουμε με διαφορετικό τρόπο. Μιλούμε για ανθρωπιστικό χώρο και θα πρέπει να μιλήσουμε και για ελευθερία δράσης των στρατιωτικών. Θα πρέπει να βρούμε τρόπο και να σεβόμαστε την ελευθερία δράσης των στρατιωτικών αλλά και το σεβασμό του ανθρωπιστικού σκέλους. Και μόνο αν τα καταφέρουμε θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο. Και καφιέμαι και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, αλλά είναι αληθές ότι με κάνει περήφανο αυτό που συμβαίνει στο Τσάντα. Στο Τσάντ λοιπόν βρήκαμε ένα μηχανισμό εργασίας, τον οποίο αναγνώρισαν πραγματικά οι συντονιστές ανθρωπιστικής βοήθειας εκείνη την εποχή. Μπορέσαμε να έχουμε μια αλληλοεκτίμηση μεταξύ των λειτουργών ανθρωπιστικής βοήθειας και των στρατιωτικών. Μπορέσαμε να έχουμε μια μέθοδο εργασίας που οικοδόμησε την εμπιστοσύνη μεταξύ ημών και ημών σεβόμενοι και τηρούμε, τηρώντας πλήρους τις αρχές. Βεβαίως δεν είμαστε ε, στο πλαίσιο της ε, προστασίας ε, του αναμάχου πληθυσμού. Θα ήθελα να πω επίσης ότι από τη στιγμή που δεν είναι καθαρά επιχειρησιακό το πρόβλημα, οι, οι, σχέσεις μεταξύ του πολιτικού και του στρατιωτικού σκέλους είναι δύσκολες, διότι είναι δύσκολο να βρεθεί ένας μηχανισμός συμφωνίας. Υπάρχουν προκαταλήψεις, στερεότυπα και είναι δύσκολο αυτό να ε, εξαφανιστεί γιατί εντάσσεται στον τομέα της ψυχολογίας. Παραδείγματα είναι το PRT στο Αφγανιστάν. Και λυπούμε διότι ο Διευθυντής Κούντς δεν είναι εδώ γιατί δεν θα με διέψευτε, αλλά στο Τσάντ δυσκολεύθηκα πολύ περισσότερο με τα στελέχη της ΕΚΟ και της ε, ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρά ε, με διάφορα στελέχη των μη κυβερνητικών οργανώσεων που είναι πολύ μακριά από το στρατιωτικό κομμάτι. Ένα άλλο πρόβλημα είναι η στρατικοποίηση της ανθρωπιστικής δράσης. Θα ήθελα να πω ότι όταν ήμουν στο γαλλικό ε, στρατό, ακόμα και ο ίδιος ο Υπουργός δεν ε, υιοθετούσε αυτή τη διατύπωση. Εγώ νομίζω όμως ότι είναι κάτι το αναπτύσσεται και το λέω διότι θεωρώ ότι πρέπει να λάβετε υπόψη σας την κοινή γνώμη. Για την κοινή γνώμη λοιπόν είναι, υπάρχει υποχρέωση, είναι προφανές ότι θα πρέπει η στρατιωτική δράση να συνοδεύεται από την ανθρωπιστική δράση. Να μην υπάρχει μόνο η, μία, ε, η πρώτη χωριστή δεύτερη. Και θα ήθελα ε, σε αυτό το σημείο να αναφέρω τη διαχείριση του χρόνου. Η διαχείριση κρίσεων από τους πολιτικούς γίνεται σε διαφορετικό χρόνο από τη διαχείριση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Αυτό καταρχάς και δεύτερον η επικοινωνία, η επικοινωνιακή δουλειά. Έχουμε ε, Quick Impact Project ε, με σχέδια γρήγορου ταχαίως αντικτύπου οι δήμοι στέλνουν στρατιώτες επιτόπου, οι οικογένειες θέλουν να στείλουν εξοπλισμό, εφόδια από τη Γαλλία στις περιοχές όπου βρίσκονται οι στρατιωτικοί τους, τα πέλη της οικογένειας που είναι στο στρατό. Και ε, ε, ε, είναι ανάγκη να ενισχυθεί η επικοινωνία, να διευρυνθεί αν θέλετε αυτό το κανάλι επικοινωνίας ως προς όλα αυτά. Από εκεί και πέρα. Ειδικά σε ό,τι με αφορά αλλά από τη στιγμή που έχω εκπροσωπήσει και διεθνή δύναμη, θέλω να πω κάτι που ισχύει και για τις ε, διεθνείς δυνάμεις, για τις κρατικές δυνάμεις, κάτι που ισχύει λιγότερο για τις ε, ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας, αλλά για τις οποίες δεν γίνεται καθόλου λόγος ε, στη δημόσια συζήτηση και θα πρέπει να γίνεται περισσότερος λόγος για όλες αυτές τις εταιρείες και τους ιδιώτες φορείς. Από εκεί και πέρα, πολύ περισσότερη η κατάρτιση για την ανθρωπιστική βοήθεια γίνεται μέσα στο στρατό και πολύ λιγότερη κατάρτιση και ενημέρωση γίνεται στους κόλπους της ανθρωπιστικής βοήθειας για την ψυχολογία των στρατιωτικών, κάτι το οποίο είναι εξίσου σημαντικό. Τελευταία παρατήρηση. Θέματα αρχής τα δέχομαι. Άλλα προβλήματα όμως υπάρχουν που μας κάνουν να δυσκολευόμαστε να συνεργαστούμε. Ε, και που ενίοτε μας φέρνουν και αντιμέτωπους θα έλεγα. Πρώτον, πολύ συχνά παρουσιαζόμαστε σαν να πρέπει να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας. Εμείς δηλαδή κάθε φορά υπερασπιζόμαστε τις χύψη αρχές. Δεν θα πρέπει να λειτουργήσουμε επιθετικά, αλλά ας μην λειτουργούμε μόνο αμυντικά υπερασπιζόμενοι το οτιδήποτε. Ας βρούμε άλλους τρόπους να προωθήσουμε ε, τις αρχές μας ή τις επιδιώξεις μας ο καθένας. Και αυτό είναι μια δουλειά που πρέπει πάντοτε βεβαίως να γίνεται τα πράγματα δεν καταχωρίζονται σε στάδια χρονικά. Δεν έχουμε πρώτα την ανάδυση του προβλήματος στις αναπτυσσόμενες χώρες που πρέπει στη συνέχεια να φτάσουν στην ανάπτυξη και ούτω καθεξής. Αντίθετα, στον ίδιο χρόνο έχουμε και το επίγον και την ασφάλεια και τη στρατιωτική παρουσία και την ανθρωπιστική βοήθεια και κάνουμε ό,τι μπορούμε σε κάθε έναν από αυτούς τους τομείς. Να καταλάβουμε δηλαδή ότι δεν διαδέχονται οι καταστάσεις τη μία ή μία την άλλη, αλλά συνυπάρχουν ταυτόχρονα και θα πρέπει να τις διαχειριζόμαστε. Από εκεί και πέρα υπάρχει το θέμα της κουλτούρας, του πολιτισμού, ε, το πνεύμα ε, που διέπει τις κοινωνίες όπου δρούμε. Το ανθρωπιστικό κομμάτι δοκιμάζεται ε, στο στίβο των διαφορετικών πολιτισμών. Ήταν ο τίτλος μιας διάσκεψης ενός σεμιναρίου στο οποίο παρέστηνα πρόσφατα. δεν λαμβάνονται σωστά υπόψη, ε, ε, λαμβάνεται σωστά υπόψη η κουλτούρα του πληθυσμού από φορείς της ανθρωπιστικής δράσης και πολύ συχνά ε, εάν δεν λάβουμε υπόψη μας αυτό το σκέλος δεν θα έχουμε επιτυχία στην ε, δραστηριότητά μας. Και εδώ τώρα απευθύνομαι σε όλους αυτούς που είναι συνάδελφοί μου ε, από το ανθρωπιστικό πεδίο. Μιλούμε πολύ συχνά για τη δυτικοποίηση, δυτικοποίηση και από ε, δυτικοποίηση, ουασιγκτονιοποίηση ή από ουασιγκτονιοποίηση, αν θέλετε, της ανθρωπιστικής βοήθειας. Δεν είναι ένα πρόβλημα εικόνας επικοινωνίας, αλλά είναι ένα πρόβλημα ε, διάρθρωσης και επικοινωνίας. Και λυπούμε διότι δυστυχώς δεν είναι μαζί μας τα μέλη πια της ε, αντίστοιχης αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου της Ιορδανίας, γιατί θα είχαν πολλά να μας πούν σε αυτό το θέμα και να μας διαφωτίσουν. Ξέρετε, και εμείς δινόμαστε την ανθρωπιστική στολή πολύ συχνά και όχι μόνο τη στρατιωτική. Και το, η αρχή που μας χαρακτηρίζει είναι το do not harm, να μην ε, προκαλούμε ε, βλάβες, να μην κάνουμε κακό όσο μπορούμε. Και τέλος, θα ήθελα να πω κάτι το οποίο μπορεί να σας φανεί προκλητικό, αλλά εννοώ να το πω. Προηγουμένως είδα μια φύσα για μια θεατρική παράσταση στις Βρυξέλλες με αντικείμενο τον Άρη και την Αφροδίτη. Μπορεί μεν ε, οι στρατιωτικοί να έρχονται από το Νάρι και οι της ανθρωπιστικής βοήθειας να προέρχονται από τον πλανήτη Αφροδίτη, ωστόσο, ωστόσο και οι δύο καλούμαστε να εργαστούμε στον ίδιο πλανήτη, τη Γη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επισκόπηση αυτή και για τις εμπειρίες που μοιραστήκατε μαζί μας από τη δράση σας. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετικό και θα είναι πολύ ωφέλιμο να σας έχουμε μαζί για την υπόλοιπη συζήτηση. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε να σας παρουσιάσουμε την προοπτική της CAR International. Είμαι της Care International. Είμαι το τελευταίο πρόσωπο, το τελευταίο ομιλήτρια του πάνελ. Θα προσπαθήσω να διατηρήσω την προσοχή σας ακεραίη. Σας ευχαριστώ που μείνατε και στην αίθουσα μέχρι τέτοια ώρα. Η Care International είναι μια οργάνωση που ε, δραστηριοποιείται για την χωροταξία, για την ε, οικοδόμηση της ειρήνης και για την ανθρωπιστική βοήθεια σε 80 ε, χώρες δραστηριοποιούμαστε εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Έχουμε λοιπόν μεγάλη εμπειρία στο πλαίσιο αυτό, όπου διάφοροι φορείς ε, προσπάθησαν να δημιουργήσουν μια τέτοια συνολική προσέγγιση και κατανοούμε πολύ συγκεκριμένα ποιοι είναι οι κίνδυνοι που ελοχεύουν σε οποιαδήποτε τέτοια ε, επιχείρηση ανθρωπιστικής βοήθειας. Και εμείς καλωσορίζουμε όπως και οι υπόλοιποι ομιλητέ, αυτή τη συνολική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε καλύτερο συντονισμό μεταξύ των φορέων, προκειμένου να υπάρχει πιο μακροπρόθεσμη ειρήνη και ασφάλεια για τις περιοχές που εμπλέκονται. Αν γίνουν σεβαστοί αυτές οι εντολές και οι ρόλοι όλων των εμπλεκομένων φορέων, όπως είπαν και προηλαλήσαντες, μια τέτοια συνολική προσέγγιση μπορεί να μας βοηθήσει να πετύχουμε τους κοινού μας στόχους, που είναι η ειρήνη και η ασφάλεια ασφαλώς. Θα παραλείψω κάποια από τα στοιχεία που ήθελα να αναφέρω για να είμαι σύντομη. Θα ήθελα να πω ότι η εμπειρία μας μας έχει διδάξει ότι πολλά θέματα προκύπτουν από την εφαρμογή της συνολικής προσέγγισης και θα ήθελα κάποια από αυτά να τα θέσω και να κάνω και κάποιες συστάσεις προκειμένου αυτή η συνολική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην αντιμετωπίσει, να μην προκαλέσει κίνδυνο σε ανθρωπιστικούς φορείς και να προωθήσει την ασφάλεια και την ευημερία των κοινοτήτων αυτών στις τόσο ευάλωτες αυτές περιοχές. Θα ήθελα να σας αναφέρω κάποιες συγκεκριμένες εμπειρίες που έχουμε αντιμετωπίσει επί τόπου και κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα θα ήθελα να σας δώσω από πλευράς των συναδέλφων μου. Παραδείγματα τα οποία ακούω καθημερινά, μου τα αναφέρουν οι συνάδελφοί μου. Είναι η καθημερινή πραγματικότητα. Του να εργάζεται κανείς σε μια ανθρωπιστική οργάνωση θα πρέπει να παραδεχτώ και να ομολογήσω ότι όταν ε, ζήτησα από τους συναδέλφους να μου πούν κατά πόσο θα μπορούσα να σας αναφέρω τα συγκεκριμένα αυτά παραδείγματα, οι συνάδελφοί μου επί τόπου έδειξαν μεγάλη απροθυμία. Δεν ήθελα να μιλήσω για πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα, για το τι συμβαίνει σήμερα επιτόπου. Είναι κρίμα, κρίμα, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μια τέτοια παρουσίαση. Αλλά νομίζω ότι αυτή η αντίδραση καταδεικνύει γιατί είναι τόσο ευαίσθητο αυτό το θέμα και γιατί εμείς ε, ως ανθρωπιστικοί φορείς θα πρέπει να είμαστε τόσο προσεκτικοί σε τέτοιες ευάλωτες περιοχές για να διατηρήσουμε και τη φήμη μας και το κύρος μας εν γέννη. Η εμπειρία καταδεικνύει ότι υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι σε περίπτωση που είναι μη αρμόζουσα και μη δέουσα αυτή η προσέγγιση από πλευράς ε, πολιτικής και στρατηγικής και κοινωτικής παρέμβασης. Ακούσαμε ότι είναι θέμα ζωής και, θανάτου. Κίνδυνη ζωής και θανάτου για τους εμπλεκομένου εμπλεκομένους φορείς, για τις κοινότητες. Πραγματικός είναι και ο κίνδυνος ανδεχόμενης απόρσησης από κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο. Είναι πραγματική λοιπόν αυτή η κίνδυνη. Και να σας πω ότι η κίνδυνη αυτή όχι μόνο είναι πραγματική, αλλά και πάρα πολύ υψηλή. Και αυτό γιατί. Διάφοροι συνάδελφοι σήμερα μίλησαν για το θέμα της θεώρησης, το πώς γίνεται αντιληπτή η ανθρωπιστική φορείς. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να γίνονται αντιληπτή ως ουδέτερη φορείς παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και να θεωρείτε ότι τηρούν αυτές τις αρχές της ανθρωπιστικής βοήθειας. Και αυτό σε μια κατάσταση όπου τα σύνορα και τα όρια μεταξύ ανθρωπιστικής πολιτικής και στρατιωτικής δράσης είναι πάρα πολύ ασαφή. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, να μένουμε και να τηρούμε τα πλαίσια της εντολής μας και να σας δείξω, να αναφέρω δύο παραδείγματα για το πώς μπορούν να λιωθούν τα όρια μεταξύ των εντολών. Ακούσαμε τέτοια θέματα σήμερα, δεν θα ήθελα να επεκταθώ από αυτού. Αλλά να αναφέρω λοιπόν ένα παράδειγμα. Όταν οι πολιτικοί φορείς παρέχουν οικονομική ε, ενίσχυση σε πολιτικές ε, ομάδες μέσω ανθρωπιστικές ε, βοήθειας. Για παράδειγμα, μια πολιτική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών ακόμα και σήμερα. Μια στρατηγική λοιπόν σε περιβάλλοντα συγκρούσεων είναι να δώσουν υποστήριξη στις δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Αυτό μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πολιτικό εργαλείο, αλλά όταν λαμβάνει τη μορφή ανθρωπιστικής βοήθειας, βοήθεια που δεν εφαρμόζεται καν βάση των ανθρωπιστικών αρχών, μπορεί να επηρεάσει την αντίληψη και τη θεώρηση των ανθρωπιστικών ε, φορέων. Αυτό αποτελεί λοιπόν ένα σημαντικό ζήτημα. Δεν έχω κάποια εξαιρετική και πανέξυπνη λύση για το θέμα αυτό. Ξέρω ότι είναι ε, μια τακτική που χρησιμοποιείται, αλλά δεν είναι σαφής. Ένα άλλο παράδειγμα και κλείνουμε αυτό είναι όταν οι πολιτικές στρατιωτικές ατζέντα σχετίζονται και συνδέονται με, το, με την χρηματοδότηση της ανθρωπιστικής βοήθειας από πλευρά μη κυβερνητικών οργανώσεων. Αυτό είναι πολύ κρίσιμη σημασία γιατί σε άλλα περιβάλλοντα οι δωρητέ άσκησαν πίεση στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις για να συνάδουν με την στρατιωτική τους και πολιτική τους ατζέντα. Σουδάν, Αφγανιστάν. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα στο Αφγανιστάν αλλά και σε άλλα και σε άλλες χώρες όπου οι δωρητές παρότριναν τις μη κυβερνητικέ ε, οργανώσεις να αναλάβουν δράση για στρατιωτικούς σκοπούς. Η ΚΕΡ, η οργάνωσή μας, δεν αποδέχεται τέτοια χρηματοδότηση, αλλά άλλες οργανώσεις αποδέχονται τέτοιες εντολές στο Αφγανιστάν, για παράδειγμα, αυτό βλάπτει όχι μόνο τη συγκεκριμένη οργάνωση, αλλά και τη φήμη όλων των μη κυβερνητικών οργανώσεων και ε, αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλειά μας και σε άλλες περιστάσεις οι δωρητέ και κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τέτοιες περιστάσεις ζητούν από τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και το έργο τους να συνάδει με τον πολιτικό του στόχο η ΚΕΡ χρειάζεται ασφαλώς χρηματοδότηση για να εξασφαλίσει την ουδατερότητά της αλλά και την ε, δυνατότητα ανάληψης δράσης της. Βλέπω ότι έχω εξατλήσει το χρονικό μου όριο. Άρα οι πιο πολλές από τις συστάσεις που ήθελα να αναφέρω έχουν ήδη αναφερθεί. Αλλά να επαναλάβω, ε, σεβασμό των ανθρωπιστικών αρχών και στην πράξη και στην πολιτική. Πρόκειται για καταστάσεις ζωής και θανάτου και για τους ε, εργαζόμενους των ανθρωπιστικών οργανώσεων, αλλά και για τα άτομα που χρειάζονται τη βοήθειά μας. Διαβούλευση με τις ανθρωπιστικές οργανώσεις, να υπάρχει διάλογος, να υπάρχει επικοινωνία. και σε ό,τι αφορά την κοινή ανακοίνωση για την ε, συνολική προσέγγιση. Υπάρχει αναφορά της ε, κοινωνίας των πολιτών, αλλά όχι συγκεκριμένα. Δεν αναφέρεται συγκεκριμένα πώς αυτό μπορεί να γίνει συστηματικά και αποτελεσματικά. Και τέλος, συνεκτικότητα της πολιτικής σε ό,τι αφορά τη συνολική αυτή προσέγγιση και αυτή η αρχή του σεβασμού των ε, ανθρωπιστικών αρχών θα πρέπει να ισχύει και για τις ευρωπαϊκούς ε, θεσμούς αλλά και για τα κράτη-μέλη. Να σας διαβεβαιώσω ότι αυτό δεν εφαρμόζεται απαραίτητα σήμερα από όλα τα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους τρεις καλεσμένους μας. Έχουμε μία ερώτηση από τον κύριο Γκέρενς και μια σύντομη θα υποβάλω και εγώ. Ευχαριστώ. Σίγουρα ήταν πολύ σύντομη αυτή η συζήτηση. Είναι πολύ σύντομη. Μακάρι να είχαμε χρόνο να τη συνεχίσουμε. Γιατί έχουν, είχαν πολύ πάθος και οι τρεις ομιλητές. Είστε κάπως προκλητικός. Το είχα καταλάβει και πριν μας το ανακοινώσετε κύριε Γανάσια. Πιστεύω ότι θα πρέπει ε, να, είμαστε, να δείξουμε κατανόηση απέναντι στην ΕΚΟ. Γιατί άλλα προβλήματα έχει η ΕΚΟ και άλλη Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού. Γιατί είναι γνωστή η φήμη του Ερυθρού Σταυρού. Είναι γνωστός ως οργάνωση, ως ε, θεσμός ουδέτερος, αμερόληπτος και οι πόρτες είναι ανοιχτές για οργανώσεις και οργανισμούς που έχουν τέτοια φήμη. Η ΕΚΟ όμω είναι ένα νέο ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο που δεν έχει χτίσει ακόμη τη φήμη τη. Και, και με την MSF είχα επαφέ και με την ΕΚΟ στη διάρκεια τη πολιτική μου σταδιοδρομία. Η MSF έχει είναι ακόμη πιο δύσκολη γιατί μερικέ φορέ αρνήθηκε χρηματοδότηση. Ε, από για χώρες οι οποίες λαμβάνουν και στρατιωτική βοήθεια, ενώ η ΕΚΟ δεν έχει τέτοιες υπερβολικές ευαισθησίες. Φυσικά και η ΕΚΟ θέλει να επιβεβαιώσει την, τη φήμη της ε, στη διάρκεια της ε, εντολής της και πιστεύω ότι έχει καταφέρει. Και από αυτή την άποψη έχει καταφέρει στις ζώνες που έχει ενεργοποιηθεί ε, να εδραιώσει τη φήμη της και νομίζω ότι χρήση αναγνώρισης. Ποιο είναι το δράμα, ποια είναι η τραγωδία των στρατιωτικών. Αποστέλλονται σε α, επιχειρήσεις ε, για να γίνουν μισητοί, ενώ οι εργαζόμενοι στον ανθρωπιστικό κλάδο ε, πηγαίνουν για να γίνουν αγαπητοί. Ενώ όλοι έχουν δικαίωμα σε αναγνώριση, γιατί το έργο και των μεν και των δε είναι απαραίτητο. Αλλά δεν θα πρέπει να συγχαίουμε τα δύο παιδεία. Σας είπα, εγώ ήμουν και υπουργό ε, ε, συνεργασίας και υπουργό ε, άμυνας και ταυτόχρονα μάλιστα. Και εκεί διαπίστωσα, έχοντας διπλή ιδιότητα, ότι πρέπει να γίνει σαφής διαχωρισμός μεταξύ των δύο. Βέβαια, μερικές φορές όταν πρέπει να σωθούν ζωές δεν θα πρέπει να εμείνουμε αμετάκλητα στο διαχωρισμό. Αλλά καταλαβαίνω γιατί με νύχια και με δόντια υπερασπίζονται και δίνουν μάχη για, το, για την ουδετερότητα και την αμεροληψία του οι εργαζόμενοι στον ανθρωπιστικό κλάδο. Συναρπαστική συζήτηση και ε, ήταν πολύ συμπαθητικά και προκλητικά τα σχόλιά σας. Μια στιγμή κύριε αν μου επιτρέπετε. Μια σύντομη ερώτηση θέλω και εγώ να υποβάλω πριν ξαναδώσω το λόγο. Όπως είπατε, στην πράξη πολύ συχνά υπάρχουν προβλήματα μεταξύ της ανθρωπιστικής και της στρατιωτικής βοήθειας. Και δεν υπάρχει μηχανισμός και ίσως και δεν χρειάζεται να υπάρχει τέτοιος μηχανισμός. Πώς όμως προσπαθούμε να λύσουμε τέτοια προβλήματα, τέτοια όπως είχαμε στο Αφγανιστάν μεταξύ στρατιωτικής και ανθρωπιστικής βοήθειας. Θα πρέπει στην πράξη να λαμβάνονται αστραπία αποφάσεις και πώς λύνονται προβλήματα όταν υπάρχει σύγχυση μεταξύ των δύο ειδών βοήθειας, της στρατιωτικής και της ανθρωπιστικής. Έχετε ένα δίλεπτο καθένας για τις απαντήσεις και για την πρόταση κάποιων λύσεων ή άντληση κάποιων συμπερασμάτων. Ο κύριος Καράσεο. Ελπίζω να μην ε, έδωσα την εντύπωση ότι ήμουν υπέρ της, ε, του συνδυασμού των δύο δράσεων, ε, η σύγχυση των δύο δράσεων. Όχι, εγώ σέβομαι αυτόν τον διαχωρισμό, γιατί έτσι ο καθένας μπόρεσε να προασπίσει και να δρεώσει τη θέση του και την φήμη του. Πολύ σημαντική δική σας ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Θα είναι κάπως ομοία απάντησή μου, υπερβολική ίσως. Εγώ δεν αυτό στο Αφγανιστάν. Εκεί ήταν η δράση αντεξέγερσης. Εκεί ο πολιτικός στόχος ήταν ουσιαστικός. Εγώ γνωρίζω καλύτερα τι ειρηνευτικές επιχειρήσει προστασία του αμάχου πληθυσμού. Εκεί ο πολιτικός στόχο είναι διαφορετικός. Και εκεί η απάντηση μου, η πρότασή μου είναι κάντε ό,τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ό,τι έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την UFOR. Μη δίνετε δράσεις στο στρατιωτικό τομέα για να ε, διενεργήσει ανθρωπιστικές δράσεις, γιατί ο καθένας θα πρέπει το έργο του να επιτελεί. Οι στρατιωτικοί να εξασφαλίζουν την ασφάλεια, αυτό είχα πει στους ε, εμπειρογνώμονες του ΣΥΜΙΚ, που μερικές φορές εκνευρίζονταν αυτό, είπα ότι εμείς είμαστε επιφορτισμένοι με την ασφάλεια. Ας αφήσουμε την ανθρωπιστική βοήθεια στους άλλους και όλο καθένας κάνει το δικό του έργο, ε, θα είναι ικανοποιημένο και ο τοπικό πληθυσμό. Γιατί δεν περιμένουν ανθρωπιστική βοήθεια από του στρατιωτικού, περιμένουν προστασία και ασφάλεια από του στρατιωτικού. Και θα πρέπει να φροντίσουμε να το λάβουμε αυτό υπόψη, γιατί τέτοια αντίστοιχη περίπτωση θα έχουμε και εντό ολίγου και στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Κύριε κυρία Μία. Uh, Νομίζω ότι ανέφερα ήδη όσα ήθελα να πω για το τι θα πρέπει να συμβεί σε ό,τι αφορά την αποφυγή της αλλίωσης των ορίων μεταξύ της πολιτικής, ανθρωπιστικής και στρατιωτικής δράσης. Νομίζω ότι πολλοί ανέφεραν σήμερα ότι κάθε φορέας θα πρέπει να περιοριστεί στην εντολή του σε ό,τι αφορά και την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, σε ό,τι αφορά την πραγματικότητα, σε ό,τι αφορά την αντίληψη του κόσμου για την πραγματικότητα και το ανέφερα εντάχει στο τέλος της σύντομης παρουσιασής μου την ανάγκη για συντονισμό και μάλιστα δομημένο συντονισμό και θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι οι φορείς επιτόπου βρίσκονται σε μια διαδικασία διαλόγου και πιστεύω πραγματικά ότι αυτό αποτελεί ένα μεγάλο τμήμα του προβλήματος, της επίλυσης του προβλήματος. Αυτό θα πρέπει να γίνει λοιπόν. Δεν είναι δυνατόν να αποστέλει κανείς ένα στρατιωτικό κομβόι ε, σε ένα ανθρωπιστικό γραφείο και να θεωρήσει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με την υπόλοιπη κοινότητα. Αυτό είναι λίγο ακραίο παράδειγμα, αλλά με το σωστό τρόπο ο διάλογος και ο συντονισμός μπορούν να βοηθήσουν να επιληθούν πολλά από τα ζητήματα αυτά. Σας ευχαριστώ και ο τελευταίος ομιλητή μας. Σας ευχαριστώ σε ό,τι αφορά το ερώτημα που θέσατε για το Αφγανιστάν. Νομίζω ότι η πρώτη απόκριση και η πρώτη ανταπόκριση θα ήταν ένας πολύ πραγματικός και αντικειμενικός διάλογος. Όπου υπάρχει πρόβλημα αλληλεπικάλυψης με το, στρατιωτικό στρατό, τι κάνουμε. Επειδή έχουμε καλό διάλογο με, τους διάφορες, τα διάφορα στρατηγία, πηγαίνουμε στο στρατηγείο, εξηγούμε το πρόβλημά μας και συνήθως επιδεικνύουν ανεκτή στάση. Φυσικά υπάρχουν περιορισμοί. Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τα πάντα, δυστυχώς. Είναι ρεαλιστική η προσέγγιση. Αν θέλουν βοήθεια, μας λένε ότι εντάξει, αλλά δεν είναι δυνατόν να προκληθεί μεγαλύτερη σύγχυση. Αν για παράδειγμα το ιδρυτικό προσωπικό ε, μεταβαίνει σε χωριά με το σήμα του Ερθρού Σταυρού μας λένε ότι κοιτάξτε, φροντίστε να υπάρχει επακριβής πληροφόρηση και από τις ερμηνείς και από την... να διευκρινιστεί ότι είσαστε προσωπικό του Ερθρού Σταυρού. Αντιμετωπίζουμε λοιπόν τέτοια θέματα και συχνά λοιπόν βρίσκουμε ρεαλιστικές και πραγματικές λύσεις για τα προβλήματα επιτόπου. Να πούμε ότι υπάρχει επίσης συμπληρωματικότητα σε κάποιες περιπτώσεις ο στρατός είναι ο μόνος που έχει τη δυνατότητα να αποκριθεί. Τα πράγματα είναι πολύ πιο περίπλοκα πάντα σε καταστάσεις σύγκρουσης. Τα πράγματα είναι λίγο πιο απλά, αν θέλετε, σε περίπτωση φυσικής καταστροφής. Αλλά η απάντηση είναι διάλογος και ρεαλισμούς. Okay. Uh, thank you uh, Καλώς. Ευχαριστώ πολύ και τους τρεις ομιλητές. και τα μέλη της Γραμματείας της Επιτροπής μας, αλλά και όλους εσάς, οι οποίοι μείνατε μέχρι το τέλος της συζήτησής μας. Νομίζω ότι ως Επιτροπή Κοινοβουλευτική Μάθαμε πολλά, καταλάβαμε πολύ περισσότερα για όλο αυτό το θέμα της ανθρωπιστικής βοήθειας, της πολιτικής βοήθειας, της στρατιωτικής βοήθειας, το πώς συνδέονται όλα αυτά μεταξύ τους. Και ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Ανάπτυξη, λοιπόν, θα πρέπει να στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις τις αρχές της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ανταλλαγή απόψεων. Ήταν απαραίτητη για εμάς για να εμπλουτίσουμε τη, γνώση μας επί του θέματος. Σας ευχαριστώ όλους. Θέλω και εγώ να επαναλάβω τα λόγια της Επιτρόπου κυρίας Γεωργίευα. Σήμερα ήταν μια πολύ καλή μέρα για την ανθρωπιστική βοήθεια. Ευχαριστώ.